Right, if if, if, if everybody could sit down, that would be very helpful, please. And then we can, we can proceed. Καθίστε παρακαλώ. Και μπορούμε να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας, αν θέλετε. Πού είναι το σφυρί μου, λέει η Πρόεδρος. Thank you. Could, could everybody sit down, please? Μπορείτε να καθίσετε παρακαλώ όλοι γιατί θα ξεκινήσει η συνεδρίασή μας. Θα ήθελα καταρχήν να συζητήσω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεύτερο σημείο ανακοινώσει της Προέδρου είναι πάρα πολύ απλές. Τα είχαμε πει και τη Δευτέρα στην τελευταία μας συνεδρίαση. Έχουμε τη μεγάλη χαρά ο Επίτροπος Μπαρνιέ, ο οποίος έχει ήδη λάβει την έγκριση των προτάσεών του από την Κομισιόν θα μας τις παρουσιάσει εδώ στην Επιτροπή μας την πρώτη ευκαιρία που υπάρχει. Είναι οι οδηγίες για την ε, αγορά των παραγών και την ανοιχτή πώληση. Απλώς λοιπόν θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο Πίτροπο να παρουσιάσει τις αποφάσεις αυτές. Της Κομισιόν δεν έχουμε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων αλλά χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία και έχουμε πραγματικά ένα προηγούμενο να μπορεί ο κύριος Επίτροπος να μας κάνει με την πρώτη ευκαιρία την παρουσίαση των ε, εξελίξεων στην Κομισιόν. Δίνω το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο, τον κύριο Μπαρνιέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και, όλ, σε όλους και όλες. Δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον της Επιτροπής σας, διότι το Σώμα των Επιτρόπων μόλις έκλεισε τη συνεδρίασή του ένα μεγάλο μέρος του πρωινού αφιερώθηκε σε μια συζήτηση σε βάθος σε σχέση με τα δύο σχέδια κανονισμού που αφορούσαν τη ρύθμιση των παραγόγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και επίσης την ε, ρύθμιση των ανοιχτών πωλήσεων short selling. Όπως ε, είχα δεσμευτεί ενώπιον σας 11 Ιανουαρίου, θα είμαι πάντα στην διάθεσή σας και γι' αυτό δίνω αυτό το θετικό μήνυμα από την πλευρά της Κομισιόν ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να παρουσιάζει πάντα τις προτάσεις της ενώπιον του Κοινοβουλίου με μεγάλη οκίτητα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι και η δική σας Επιτροπή εργάστηκε πολύ σκληρά για τα, τους κανονισμούς αυτούς. Το λέω αυτό γιατί αυτά τα οποία κάνετε σε όλο το θέμα, σε όλα τα θέματα της εποπτείας των χρηματαγορών και ιδίως για τα παράγωγα προϊόντα και τις ανοιχτές πωλήσει, όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα προετοιμασίας των κειμένων και βοήθησαν ιδιαίτερα την ομάδα μου, τους συνεργάτες μου και εμένα τον ίδιο. <laughs> και υπάρχει ο Ντάβιτ Ράιτ, ο, γενικός, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συμβολή του. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Μπέρνατ Λάγκεν, ο οποίος είναι παρόν από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Σομ Πολ Γκοζές για το σημαντικό ρόλο που έχουν αναλάβει σε σχέση με τα δύο αυτά σχέδια ε, κανονισμών. Και όπως είπα και στο Σώμα των Επιτρόπων, το γενικό πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα πλέον, χάρη στην πάρα πολύ επικοδομητική και ευφυά εργασία των εισηγητών σας για τα χρήματα οικονομικά και τους οποίους θέλω και πάλι να ευχαριστήσω. Και χάρη στη συμφωνία που επέτυχε η Βελγική Προεδρία στο Συμβούλιο Κόφιν έχουμε ήδη ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να εγγραφεί η επιμέρους κατά προϊόντα, κατά τομέα, κατά αγορά νομοθεσία ρύθμισης για τα χρηματοοικονομικά θέματα. Γι' αυτό οι τα νομοθετήματα αυτά για τις χρηματοοικονομικές αγορές που θα εγκρίνει ελπίζω το Κοινοβούλιο σας την επόμενη εβδομάδα είναι τελικά η αποκριστάλλωση όλων των πρωτοβουλειών που έχουμε αναλάβει για να υπάρχει σταθερότητα στις χρηματαγορές της Ευρώπης και να υπάρχει η πρέπουσα εποπτεία και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, η βασική μας φροντίδα, θέλω να το τονίσω εδώ, είναι να κινούμαστε εν παραλίλω με τους Αμερικανούς και τις άλλες περιοχές του κόσμου. Είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός να μην θέσουμε σε μειονεκτική θέση την ευρωπαϊκή οικονομία εναντί άλλων περιοχών του κόσμου, ιδίως εναντί των Ηνωμένων Μετά από την συνεδρίαση των G20 θα πρέπει το φύλλο πορείας να τεθεί σε λειτουργία, σε να υλοποιηθεί εν παραλίλω. Όχι πάντα με τα ίδια μέτρα, γιατί δεν είναι ακριβώς ταυτόσιμες οι τραπεζικές μας και χρηματοπιστωτικές μας υπηρεσίες, οι εθνικές αρχές, αλλά με παράλληλο τρόπο. Γι' αυτό έκανα μια πρόσφατη επίσκεψη στις ΗΠΑ και θα επανέλθω ως Νούπο για να διακριβώσω ακριβώς κατά πόσο υπάρχει αυτός ο παραλληλισμός στις εργασίες μας. Όπως έλεγα προηγουμένως, τα παράγωγα προϊόντα έχουν μια τεράστια οικονομική σημασία. Μιλάμε για ένα όγκο συναλλαγών που έχει αυξηθεί ραχδαία, όπως αναφέρει και ο κύριος Λάγκες στην έκθεσή του τα τελευταία χρόνια. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε 6.000 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό όγκο συναλλαγών στα παράγωγα. Η τωρινή κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική γιατί τα 80% αυτών των συναλλαγών γίνονται ε, εκτός χρηματαγορών, over the counter δηλαδή όπως λέμε, χωρίς, κανένα, χωρίς καμία δυνατότητα ελέγχου. Αυτό δεν οδηγεί σε ανακάλυψη των τιμών, οδηγεί σε μια ε, μεγάλη διακύμανση των τιμών και ευνοεί κερδοσκοπικά φαινόμενα. Γι' αυτό είναι προς το συμφέρον μας να εξασφαλίσουμε τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών παραγωγών μέσα στα πλαίσια που έθεσαν οι G20. Okay. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα στους θαλάμους διερμηνίας. Θα πρέπει να κάνουμε μισό λεπτό διάλειμμα μέχρι να μου πούνε ότι όλα δουλεύουν καλά.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 Euh, je parlais du parallélisme avec les Américains, mais aussi avec les autres régions. D'ailleurs, dans quelques jours, je rendrai public. Μιλούσαμε για τον παραλληλισμό με τι άλλε περιοχέ του κόσμου. Θα κάνουμε σε ορισμένε μέρε μία άσκηση βαθμονόμηση, συγκριτική ε, αξιολόγηση εναντί των άλλων περιοχών του κόσμου και βλέπετε ότι όλα αυτά βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας εξασφάλισης του παραλληλισμού. Το πρώτο λοιπόν αυτό κείμενο για τα παράγωγα προϊόντα τι περιλαμβάνει. Λέμε ότι η διαφάνεια δεν είναι επαρκής αυτή τη στιγμή στις χρηματαγορές. Γι' αυτό εμείς θα δώσουμε έμφαση στην ανιχνευσιμότητα των παραγωγών και των συναλλαγών παραγωγών Καταρχήν με το να ευνοήσουμε την τυποποίηση ώστε να τον περισσότερο των προϊόντων αυτών και σας πεθυμίζω ότι αν κάποια παράγωγα φαίνεται να έχουν επικίνδυνο χαρακτήρα χάρη στο Κοινοβούλιο, χάρη στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο εισηγητής σας κ. Σφεν Χίγκολτ θα υπάρχει δυνατότητα από την ρυθμιστική αρχή αγορών να απαγορεύονται αυτά τα παράγωγα. Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών θα καταγράφεται πλέον σε ειδικά μητρώα συναλλαγών, ένα είδος μαύρων κουτιών που θα κρατάνε τη μνήμη όλων των κινήσεων αυτών των ε, αξιογράφων των, στα λεγόμενα trade repositories που είναι η μνήμη της ε, κίνησης αυτών των παραγωγών. Επίσης θα ενθαρρύνουμε τον συν, τον συμψηφισμό, γιατί και αυτό είναι ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και επίση και μεγαλύτερη ασφάλεια των χρηματοοικονομικών συναλλαγών αυτών. Και φυσικά θα λαμβάνουμε υπόψη τις υποχρεώσεις ιδίου κεφαλαίου για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Όταν αυτά τα ιδρύματα ε, χρησιμοποιούν την οδό του συμψηφισμού, τότε θα είναι χαμηλότερε οι κεφαλογικέ ε, απαιτήσει για αυτά τα ιδρύματα. Θα πρέπει λοιπόν να περνάνε από κεντρικό συμψηφισμό, από ένα ίδρυμα κεντρικού συμψηφισμού και όχι μόνο από διμερή συμψηφισμό τα παράγωγα για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή μόνο 30% των παραγόγων υπόκεινται σε συμψηφισμό. Οι συναλλαγές λοιπόν που έχουν να κάνουν με swaps επιτοκίων και 10 ως 20 για, τα, ε, για τις ανταλλαγές, υποχρεω, για τις ε, ανταλλαγές υποχρεώσεων αθέτησης, τα credit swaps. Όπως όμως έχουν κάνει και οι Αμερικανοί, εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες, πολλές από αυτές, όταν εξάγουν ε, προϊόντα, χρησιμοποιούν παράγωγα για την κάλυψη κινδύνων για την αντιστάθμιση κινδύνων. Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν αυτά τα παραγωγά προϊόντα για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά αντίθετα για στόχους ε, αντιστάθμισης και προστασίας των δραστηριοτήτων που ασκούν στην Ευρώπη. Επομένως, γι' αυτό το λόγο έχουμε αποφασίσει να προτείνουμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τα παράγωγα για λόγους αντιστάθμισης δεν πρέπει να υπόκειται στις υποχρεώσεις όπως και οι χρηματοοικονομικοί εταίροι στις αγορές. Επομένως, αν το κάνουν για λόγους αντιστάθμισης, τα τη χρήση των παραγάγων δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Ενώ αν χρησιμοποιούν αυτά τα παράγωγα όπως θα κάνουν χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τότε θα υπόκειται πλήρως στους κανόνες που αφορούν και σε όλα τα ιδρύματα. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα της αγοράς ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνεται θετικά η εποπτεία και θα γίνεται ταχαίως ο συμψηφισμός των παραγωγών. Γι' αυτό οι κεντρικοί φορείς συμψηφισμού βρίσκονται στην καρδιά αυτού του συστήματος και επίσης θεωρούμε ότι η ΕΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών, είναι αυτή η οποία θα πρέπει να εποπτεύει τα trade repositories, τα μητρώα συναλλαγών και επίσης να παίζει τον απαραίτητο ρόλο για τη ρύθμιση των αγορών. Λίγα ακόμα λόγια κυρία Πρόεδρε. Προφανώ θα είμαι στη διάθεσή σα σε μια μεταγενέστερη στιγμή για να προβώ σε διάλογο μαζί σα για αυτό το θέμα που ούτω ή άλλω θα σα απασχολήσει το θέμα τη ανοιχτή πώληση, short selling. Η πώληση αξιογράφων ή στοιχείων ενεργητικού χρηματοοικονομικού χαρακτήρα με ανοιχτή πώληση όταν κανείς δεν έχει καν τη δυνατότητα ότι μπορεί να καλύψει εκ των υστέρων την ανοιχτή πώληση, αυτό είναι μια πρακτική που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς θεωρούμε, και αυτό δεν είναι μια ιδεολογική προσέγγιση, ότι η ανοιχτή πώληση, ιδίως ό,τι αφορά το κρατικό χρέος, μπορεί να έχει κάποιες θετικές πτυχές να ευνοεί την ρευστότητα, παραδείγματο χάρη. Γι' αυτό το λόγο δεν αντιμετωπίζουμε ιδεολογικά τα θέματα τη ανοιχτή πώληση, αλλά μονάχα με το στόχο να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ρύθμιση και να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στι συναλλαγέ αυτέ. Ποιε είναι οι βασικέ αρχέ λοιπόν του κειμένου μα στα θέματα αυτά. Η κάθε ανοιχτή πώληση θα πρέπει να καταγράφεται, να γίνεται το λεγόμενο flagging, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό. Όπω το κάνουν ακριβώ και οι Αμερικανοί. Αυτό είναι κάτι καινοφανέ στην Ευρώπη η ταυτοποίηση, η συστηματική ανείχνευση και ταυτοποίηση και υποχρεωτική ταυτοποίηση οποιασδήποτε ανοιχτή πώληση ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να παρακολουθήσουν την κίνηση των αγορών και μπορούν έτσι να αξιολογήσουν την αύξηση του κινδύνου ενδεχόμενα. Αυτό γίνεται και στις ΗΠΑ και στο Χονγκ Κονγκ. Επίσης μας ενδιαφέρει η διαφάνεια κάθε φορά που ένας φορέας της αγοράς ε, θέτει σε πώληση ένα σημαντικό όγκο αξιογράφων μιας επιχείρησης ή ενός κράτους θα πρέπει να το δηλώνει. Αν πουλιέται πάνω από 0,2 του κεφαλαίου μιας επιχείρησης θα πρέπει αυτό να αναφερθεί στις ρυθμιστικές αρχές. Επίσης, αν ξεπερνάμε το 0,5% στην αγορά πάλι θα πρέπει να ισχύουν αντίστοιχες υποχρεώσεις για το χρέος των ε, κρατικών, το κρατικού χαρακτήρα. Επομένως, οι ανοιχτέ πωλήσει θα πρέπει να ελέγχονται για να εξασφαλίσουμε ότι κάποιος ο οποίος προβαίνει σε ανοιχτή πώληση έχει πράγματι τη δυνατότητα να καλύψει τη θέση του είτε με αγορά τίτλων είτε με δανεισμό. Εάν δεν υπάρξει αυτή η προφύλαξη και αν κάποιος δεν είναι σε θέση να παραδώσει τους τίτλους τους οποίους έχει αποκτήσει με ανοιχτή πώληση, τότε την τρίτη μέρα θα είναι υποχρεωμένος να σταθεροποιήσει την θέση του και εάν δεν το πράξει θα υποστεί κυρώσεις από τη ρυθμιστική αρχή. Αυτό είναι μια νέα λοιπόν αρχή η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ε, ε, ενίας αγοράς. Είναι μια προσέγγιση παράλληλη με αυτή που ακολουθείται στις ΗΠΑ. Εμείς δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε τι ανοιχτέ πωλήσει, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα για τι πράξει αυτέ. Πιστεύω λοιπόν κυρία Πρόεδρε ότι με αυτού του δύο σημαντικού κανονισμού που έχουν υποστηριχθεί και από τον φίλο και συνάδελφο Όλη Ρεν, ο οποίο έχει υποστηρίξει όλο το πακέτο τη εποπτεία σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου στο παρελθόν. Για... Χάρη σε όλα αυτά τα νομοθετήματα δεν είμαστε πια τόσο απροστάτευτοι όσο ήμασταν στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών κρίσεων και θα εργαστούμε όπως έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ πιο ευρωπαϊκό από ό,τι στο παρελθόν δίνοντας σε ανεξάρτητες αρχές των αγορών και στην ΕΣΜΑ τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα συντονισμού των δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίω για τι ανοιχτέ πωλήσει, με μηχανισμούς εναρμονισμένους, λήψεις αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών και με εναρμονισμένους μηχανισμούς συντονισμού για την αγορά, για την Επιτροπή, για την Αρχή Ρυθμιστική Αγορά, ε, Επιτροπή Αγορών, η οποία να, να είναι, ε, δρά 24 ώρες το 24 ώρο. Όλα αυτά τα κείμενα λοιπόν έτυχαν επεξεργασία στι τελευταίε εβδομάδε και πρέπει να σα πω και πάλι ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμε και επικοδομητικέ οι συμβολέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, το θέμα προηγουμένω σε σχέση με τον απαραίτητο χρόνο για να μπορέσουν να τεθούν εν εφαρμογή όλοι αυτοί οι κανονισμοί. Υπάρχει ένα τεχνικό χρόνο που χρειάζεται, που μπορούμε πάντα να τον μειώσουμε, αλλά υπάρχει και ο χρόνο ο δημοκρατικό κατά κάποιο τρόπο για τη λήψη αποφάσεων. Αυτό εξαρτάται και από εσά και από το Συμβούλιο και εδώ θα πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα και θα ελπίσω θα θέλω να ελπίζω ότι εσείς μπορείτε να καθορίσετε τους εισηγητές σας τάχει ώστε τα δύο αυτά πακέτα ρύθμισης να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατό και από τα δύο νομοθετικά σώματα. Οι υπηρεσίε μου είναι στη διάθεσή σας και τις επόμενες εβδομάδες σε σχέση με τα, τα μία επίλυσης και για τους ε, ε, φορείς αξιολόγησης και για άλλα νομοθετήματα όπου εγώ έχω προτείνει να υπάρξει σημαντική ε, ενίσχυση του καθεστώτος κυρώσεων, όλες αυτές οι οδηγίες από κοινού θα βοηθήσουν να έχουμε ένα πληρέστερο πλαίσιο εποπτείας το οποίο θέλουμε να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Commissioner. Um, σας ευχαριστούμε πολύ. Εκτιμούμε το γεγονός ότι ήρθατε εδώ να μας ε, ενημερώσετε, να μας κάνετε αυτήν την εισήγηση όσο γινόταν πιο έγκαιρα. Και βεβαίως ε, η Επιτροπή μας ε, αδειμονεί να μάθει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής. Είμαι βέβαια, όπω θα θυμάστε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του πακέτου για την εποπτεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να συνεργαστούμε. Και πιστεύω πως αυτές οι προτάσεις σε κάποιο βαθμό θα το δοκιμάσουν αυτό αμέσως. Όπως αναγνωρίζετε για το ρόλο της ε, τραπεζικής αρχής ε, στη δημιουργία απαιτήσεων για τους βασικούς εταίρους. Αλλά βεβαίως θα υπάρξουν και άλλες επιδράσεις στον τραπεζικό χώρο που έχουν να κάνουν με την κοινοποίηση πληροφοριών. Με βέβαια ότι οι συνάδελφοι θα τα δούμε όλα αυτά όταν θα μπούμε στις λεπτομέρειες των προτάσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα θέλαμε να σας ξαναδούμε σύντομα. Um, Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στην ακρόαση για τη βελτίωση της οικονομικής ε, διακυβέρνησης και το πλαίσιο σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα της ζώνης του ευρώ. Να καλωσορίσω τους ομιλητές μας για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον ε, της ε, διάρθρωση, ε, μιας διαδρομένη μάλλον διακυβέρνηση τη Ένωση. Ε, είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση αυτή, γιατί υπάρχουν πολλέ δραστηριότητε που θα γίνουν σχετικά στι επόμενε εβδομάδε. Ε, οι Υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν ήδη. Αύριο ο πρόεδρο Φανορών Πάη θα δώσει προφορική ενημέρωση για τη συνέχιση των εργασιών τη Task Force και στα τέλη του μήνα η Κομισιόν θα δώσει τι προτάσει τη για το νέο πλαίσιο οικονομική διακυβέρνηση κυβέρνησης. Επίσης, στη δική μας Επιτροπή θα συζητήσουμε τις τροπολογίες στην έκθεση ΦΕΡ για τις 27 Σεπτεμβρίου με ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, στις 24 Οκτωβρίου ώστε να εγκριθεί στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Όλοι δουλεύουμε σκληρά λοιπόν ε, και βλέπουμε να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Επίκαιρη λοιπόν η σημερινή μας ακρόαση. Καταρχήν θα έχουμε την ευκαιρία για μια ανταλλαγή απόψεων με τον Λορέντζο Σμάγκη που είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με τον Επίτροπο Όλη Ρεν που δεν χρειάζεται καν να σας το συστήσω. Στη δεύτερο τμήμα θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον πάνελιστ Κάρλο Κοτορέλη, Στεφάν Κονιλινιόν και Αντρέ Σαπιέ θα ισχύσει η αρχή του Catch the Eye για τον χρόνο αγόρευσης των μελών και θα πρέπει να σας θυμίσω σε όλους ότι πρέπει να τελειώσουμε αυτήν εδώ τη συνεδρίαση στις 18 ε, και 15, δηλαδή 6 και 4. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι τις 6.30 διότι ξεκινήσαμε νωρίτερα. Και ζητώ συγγνώμη διότι θα πρέπει να εγκαταλείψω την Προεδρία λίγο πριν από το τέλος γιατί ξεκινάει ένας τριμερής διάλογος. να στραφώ στον πρώτο μας ομιλητή, τον Λορέντζο. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σε ευχαριστώ που μου προσφέρετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σε ένα θέμα το οποίο είναι τόσο επίκαιρο όσο και ιδιαίτερα σημαντικό επίκαιρο, διότι σε λίγες μόνο εβδομάδες η Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει τις νομοθετικές της προτάσεις και ο κύριος Φαν Ρόμπεϊ θα παρουσιάσει σε ένα μήνα την έκθεση για την ομάδα κρούσης που έχει συστήσει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αποδείξουμε ότι επίγει να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση και το πλαίσιο σταθερότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Ευρωζώνης. Για να βελτιώσουμε λοιπόν τη διακυβέρνηση και, την, και το πλαίσιο πλαίσιο σταθερότητα ε, της Ευρωζώνη, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι δεν πήγε καλά με το προηγούμενο σύστημα και η κίνδυνη που συνεπάγεται η αποτυχία εάν ε, αυτή επαναληφθεί. Ε, Νομίζω οι περισσότεροι συμφωνούν τώρα για το τι δεν πήγε καλά. Το σύστημα δεν ήταν σε θέση να επιβάλλει πειθαρχία, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο σε μια νομισματική ένωση. Πιο συγκεκριμένα, οι μηχανισμοί σχεδιασμένοι για την πειθαρχική, ε, δημοσιονομική πειθαρχία δεν λειτουργήσαν ε, όπως αναμενόταν. Ε, δεν ε, περίμενε κανείς ότι θα υπάρξει τόσο μεγάλο χρέος και όταν προέκυψε αυτό δεν ε, λάβαν χώρα ε, ταχύτατα οι απαραίτητες διορθώσεις. Κατόπιν οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν λειτουργήσαν ως αποτρεπτικό μέσο και κατόπιν τούτου είχαμε ένα συνδυασμό μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, της χειρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Αφενό και αφετέρου τη σώρευση ανισορροπιών στην Ευρωζώνη, κάτι το οποίο οδήγησε στο να μην δοθεί απαραίτητη προσεχή στην ανταγωνιστικότητα και στι ε, απαράδεκτε δημοσιονομικέ πολιτικέ. αυτό το μείγμα ήταν ένα πολύ μεγάλο βάρος για πολλές χώρες. Οι χώρες της ε, Ευρωζώνης δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νομισματικά εργαλεία για να, πληθω... να πληθωρήσουν το ε, χρέος. Κάτι, να του δώσουν μια νομισματική μάλλον χρειά, όπως έγινε πριν από 10 περίπου χρόνια. Το πρώτο θέμα που παίζει ρόλο είναι ότι οι ίδιες οι χώρες, οι χώρες έχουν και προβλήματα να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. Θεωρείται ότι αυτό δεν είναι και πολύ σημαντικό για το Σύμφωνο σταθερότητα, είχε ως στόχο ακριβώ να αποτρέψει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο θέμα είναι ότι οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ μπορούν ταχύτατα να αλλάξουν γνώμη για την φερεγγιότητα μια χώρας και με τον τρόπο αυτό προκαλούν εξελίξεις. Το γεγονός ότι μπορεί κανείς να κερδίσει χρήματα από τη χρεοκοπία μιας εταιρείας ή ακόμα και μιας χώρας χωρίς να έχει κάνει καμία απολύτως επένδυση, αυτό βεβαίως θίγει το θέμα της λειτουργίας των χρηματοψηφικών αγορών, κάτι το οποίο μέχρι πριν από λίγο δεν εξετάσαμε. Και ε, νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτη η ανακοίνηση Κομισιόν επί του θέματος. Το τρίτο πρόβλημα είναι ότι ε, μια ε, χρεοκοπία κρατική έχει άμεσες επιπτώσεις και γι' αυτό λοιπόν οι κίνδυνοι που συνδέονται με ένα μικρό κομμάτι της Ευρωζώνης είχαν τόσο σημαντικές επιπτώσεις στο ευρώ. Η τρίτη αυτή διάσταση ακόμα δεν έχει γίνει πλήρω κατανοητή, παρότι είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία έχοντα κατά νου τις αλλαγές που πρέπει να λάβουν χώρα στη θεσμική δομή τη Ευρωζώνη. Η αλληλένδεση ανάμεσα στα διάφορα νομίσματα τροποποίησε αυτό που κατά την άποψή μου ήταν ένα περιορισμένο πρόβλημα ή το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας η το προβλημα τη ελληνική οικονομία, κάτω από 3% του ε, ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμω, το μικρό πρόβλημα μετατράπηκε σε συστημικό και γι' αυτό εξηγεί ότι όταν οι αγορές άρχισαν να αμφιβάλλουν για την φαραγγιότητα της Ελλάδας ξεκίνησαν ε, κερδοσκοπικές κινήσεις οι οποίες επηρέασαν και άλλες χώρες και ε, δημόσια οικονομικά στην ίδια την Ευρωζώνη. Προκέπτυψε λοιπόν ένταση και φτάσαμε ε, σε πολύ μεγάλη σε επίπεδο ένταση σε πάρα πολλού τομεί. Ε, Μερικέ φορέ μάλιστα ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ακόμα και από αυτή που διαπιστώθηκε αμέσω μετά την αποτυχία τη ε, Τράπεζα Lehman Brothers. Δεν θα αναφερθώ ε, σε αυτά, αλλά μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο που σα έχω δώσει κάποια στοιχεία, δείκτε για το... Διακόπτω τον ομιλητή, γιατί μιλάει με απίθανη ταχύτητα βέβαια και θα προσπαθήσω λέει να μιλάω λίγο πιο αργά. Ευχαριστούμε πολύ. Ε... Ε, στο έγγραφο λοιπόν που σας έχω δώσει ε, φαίνεται πόσο οξία ήταν αυτή η κρίση και οι κίνδυνοι ε, που έλαβαν χώρα εμφανίστηκαν στην Ευρωζώνη. Σε γενικές λοιπόν γραμμές το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου το παγκόσμιο δημοσιονομικό σύστημα ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. βέβαια σας είπα, ε, ήταν και ακόμα χειρότερα από ό,τι συνέβη μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. Ε, ε, ε, θα είχαν καταρρεύσει οι αγορές αν δεν συμφωνούσαμε εμείς να συστήσουμε ένα ταμείο σταθερότητας που θα βοηθάει τις χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο και αν δεν είχε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει άμεσα σε ορισμένες αγορές για να επαναφέρει την εύρυθμη λειτουργία τους. Έτσι λοιπόν οι μετέχοντες στην αγορά οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί βραχυπρόθεσμα απέναντι στο ευρώ και απέναντι σε κάποια δημόσια κεβάλαια αυτοί υπέστησαν ζημιές και έτσι διατηρήθηκε η ακαιρεότητα της Ευρωζώνης. Θα ήταν βέβαια λάθος να πιστέψουμε ότι οι κίνδυνοι που εμφανίστηκαν την Άνοιξη δεν θα εμφανιστούν ποτέ πια. Εάν οι αδυναμίες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της Άνοιξης δεν αντιμετωπιστούν οριστικά και αμετάκλητα, είναι αναγκαστικά, ε, μάλλον είναι ε, δυνατόν να επανέλθει η αστάθεια και ο κύριος Ρόμπαι έχει το καθήκον να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για να αποφευχθεί τέτοια κατάσταση. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να κλείσουν όλα τα παραθυράκια ε, που έχουν σχέση με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον τρόπο αυτό να μην είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτεθειμένη σε μελλοντικέ επιθέσεις. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Οποιαδήποτε αλλαγή στη θεσμική δομή της Ευρωζώνης και του Ευρώ πρέπει να ξεκινήσει με τις ίδιες απλουστευμένες παραδοχές που κάνουμε και κατά το παρελθόν και θα ήθελα εδώ να φέρω τρεις. Η πρώτη απλουστευμένη παραδοχή που κάνουν και συχνά οι οικονομολόγοι είναι να πιστεύουν ότι οι αγορές είναι πάντα σωστές ε, και μπορούν να ε, πειθαρχήσουν τις αγορές. Ξέρουμε ότι κατά το παρελθόν ίσως ε, υπήρξε λάθος αξιολόγηση στην ε, υπερτίμηση του κινδύνου και ενδέχεται κάποια στιγμή στο μέλλον να υπάρξουν διορθώσεις. Ε, το να αφήνει λοιπόν κανείς αγορές ε, το καθήκον, να, στις αγορές το καθήκον να επιβάλλουν εκείνες την πειθαρχία, αυτό είναι πάτη που μπορούν να έχουν μόνο οικονομολόγοι. Αν πραγματικά θέλουμε να προλάβουμε και να διορθώσουμε τι ισορροπίε κυρίω τι δημοσιονομικέ, χρειαζόμαστε ισχυρότερου θεσμούς, θεσμικούς μηχανισμούς στην Ευρωζώνη και στις ε, χώρες που έχουν την Ευρωζώνη. Το δεύτερο λάθος που πρέπει να αποφύγουμε είναι να πιστεύουμε ότι γενικά μπορούμε να αποφύγουμε την κρίση. Οι κρίσεις έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν και ίσως και επανεμφανιστούν στο μέλλον και για λόγους ε, μόλυνσης σε εισαγωγικά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι και να τι αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Το τρίτο λάθο είναι να πιστεύουμε ότι ε, πολύ εύκολα ε, και με τάξη βγήκαμε από την κρίση. Οι κρίσει όμω, όπω σα είπα, μπορεί να είναι μολυσματικέ και να έχουν απρόβλεπτε συνέπειε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει καταρτήσει συγκεκριμένε προτάσει για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Είναι γνωστέ οι προτάσει, έχουν κοινοποιηθεί. Εγώ θα αναφερθώ σε τρία βασικά μόνο στοιχεία που έχουν έχουν σχέση με την δημοσιονομική πειθαρχία, τη μακροοικονομική υποπτία και την διαχείριση της κρίσης. Θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο γενικής φύσεως σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι οι προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν αλλάζουν τη φύση της Ευρωζώνης, κυρίως όσον αφορά τον επιμερισμό των ευθυνών και σε σχέση με τη δημοσιονομική πολιτική η οποία παραμένει στα χέρια των εκάστοτε εθνικών αρχών. Άρα δηλαδή για μας δεν είναι απαραίτητο στην Ευρωζώνη να Υπάρχει μία και μόνο δημοσιονομική, ε, πολιτική. Ούτε είναι απαραίτητο να υπάρχει μία transfer union όπως λέγεται. Βέβαια, οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να χαράσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο που καθορίζεται από το ενιαίο νόμισμα. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στη διακυβέρνηση, την οικονομική, να ενισχύσουμε την πειθαρχία πρώτα απ' όλα για τις χώρες της Ευρωζώνης, να προβούμε σε πλήρη χρήση των ε, ρυθμίσεων της συνθήκης, κυρίως του άρθρου 136, το οποίο προσθέθηκε στη νέα συνθήκη ακριβώς διότι τα κράτη-μέλη της Νομισματικής Ένωσης πρέπει να επιδεικνύουν ακόμα καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση και οτιδήποτε αποφασίζεται για την Ευρωζώνη μπορεί βεβαίως να εφαρμόζεται και στο υπόλοιπο της Ένωσης αν αποφασιστεί έτσι. Πάντως η συζήτηση ανάμεσα στους 27 κατά την άποψή μας δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε αυτά που διαδραματίζονται στην Ευρωζώνη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο της ισχύουσας συνθήκης συνθήκης μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δευτερογενή νομοθεσία. Και δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουμε το τελευταίο τμήμα των προτάσεων τις οποίες έχουμε καταθέσει. Επίσης, να πω ότι δεν έχουμε και χρόνο δεν μπορούμε να περιμένουμε αλλαγή της συνθήκης. Όπως είπα προηγουμένως, οι αμφιβολίες που έχουν εκφράσει οι χρηματοπιστωτικές αγορές για την ικανότητα του συστήματος να είναι πιο ανεκτικό, αυτές οι αμφιβολίες πρέπει να εξαφανιστούν το συντομότερο δυνατόν. Και αν καθυστερήσουμε πάλι θα ε, διαχυθούν οι αμφιβολίες. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε συζητήσεις που έγιναν για τρία βασικά θέματα της μεταρρύθμισης. Όσον αφορά την δημοσιονομική διακυβέρνηση, το πρώτο βήμα έγινε σε 7 Σεπτεμβρίου, όταν το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ αποφάσισε για ένα νέο πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλύτερη δημοσιονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει τη δημιουργία εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων που δημιουργούν ελάχιστα προαπαιτούμενα για την συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς και στατιστικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα προάγουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία στις εθνικές δημοσιονομικές ε, αξιολογήσεις, πρότυπα υψηλής ποιότητος, μια καλύτερη μεσοπρόθεσμη προσέγγιση και καλύτερη κάλυψη όλων των δημοσιονομικών σε κυβερνητικό επίπεδο. Πέντε μέτρα λοιπόν θέλει να προωθήσει η Κεντρική Τράπεζα. Καταρχήν, πιο ταχείες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών εξέλιξεων. Δεύτερον, αναστροφή του βάρους απόδειξης, κάνοντας πιο δύσκολο για το Συμβούλιο να αλλάξει τις αποφάσεις στις αποφάσει του την αξιολόγηση κομισιών. Τρίτον, μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην συλλογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δεδομένων. Τέταρτον, μεγαλύτερη έμφαση στην παρακολούθηση του εθνικού χρέου. Και πέμπτο, σχεδόν αυτόματο χαρακτήρα των κυρώσεων σε περίπτωση παραβίαση των κανόνων. Η ανακοίνωση της Κομισιόν της 12 η Μαΐου πηγαίνει σωστή κατεύθυνση, θα θέλαμε όμως να είναι πιο φιλόδοξη σε δύο πτυχές. Πρώτον απ' όλα. Καταρχήν, μέχρι στιγμή η Κομισιόν σιωπή σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η ανεξαρτησία των δημοσιονομικών και ποιοτικών αξιολογήσεων τη στατιστική συλλογή δεδομένων μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική στην Κομισιόν την ίδια. Θα θέλαμε να δούμε κάποιε από τι διαδικασίε οι οποίε εφαρμόζονται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού σε επίπεδο τεχνικών αξιολογήσεων και το ρόλο του Επιτρόπου του Αρμόδιου να εφαρμόζεται και στην περίπτωση της ε, ΕΚΦΗΝ, της Γενικής Διεύθυνσης για τα Χρηματοοικονομικά. Σε ό,τι αφορά τις στατιστικές, ο νέος κανονισμός Συμβουλίου του Ιουλίου 2010 θα πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερους πόρους για τη Eurostat και την ε, επαλήθευση των δημοσιονομικών στοιχείων. Δεύτερον, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες και οι προτάσει Κομισιόν δεν βελτιώνουν ιδιαίτερα την κατάσταση. Ήταν πολλέ φορέ στο παρελθόν ότι είναι ιδιαίτερα επαχθεί και μακροσκελεί οι διαδικασίε μέχρι ότου να μπορεί να αναλυφθεί αποτελεσματική δράση για να υπάρχουν κίνητρα ή επιβολή μέτρων εναντίον των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τι δημοσιονομικέ του εξέλιξει. Μέχρι τώρα οι διαδικασίε έχουν ξεκινήσει μονάχα επί τη βάση κοινοποιήσεων από τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσε κανεί να φαντάζεται μια διαδικασία που να βασίζεται στην αξιολόγηση εκ των προτέρων από την Κομισιόν για τα κράτη-μέλη. Γιατί αν είχε γίνει αυτό στην περίπτωση τη Ελλάδο, πολλά προβλήματα θα είχαν αποφευθεί ή θα είχαν τουλάχιστον ε, μετριαστεί. Στο δεύτερο στοιχείο, τη μακροοικονομική εποπτεία, βλέπουμε την ανάγκη να γίνει ένα καφαντικό άλμα δεδομένη στι ε, επιπτώσει που έχουν οι μακροοικονομικέ πολιτικέ μια χώρα στι υπόλοιπε χώρε τη ζώνη του ευρώ. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτείνει, προτείνει τη δημιουργία ενό μηχανισμού επαγρύπνηση που να βασίζεται σε, μια σαφή, ε, σε ένα σαφέ σύνολο δικτών που δείχνει πότε μια πολιτική δεν είναι βιώσιμη σε οικονομικό επίπεδο. Θα θέλαμε και πάλι η Κομισιόν να δείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία και να ακολουθήσει την οδό της ε, πίεσης προς τα, προς τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν τις μακροπρόθεσμες βάσεις μιας οικονομικής ένωσης. Τρίτο στοιχείο, η διαχείριση των κρίσεων. Υπάρχει μια, καλή υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι αν έχουμε ένα καλό σύστημα πρόληψης δεν θα υπάρξουν κρίσεις. Θεωρία είναι αυτό βέβαια. Στην πράξη οι κρίσεις λαμβάνουν χώρα ακόμα και αν τα θεσμικά, τα θεσμικά συστήματα για την εποπτεία και την πρόληψη είναι αρκετά ισχυρά. Θα ήταν λάθος όπως είπα προηγουμένως, αλλά θα ήταν και ανεύθυνο να θεωρούμε ότι δεν θα επαναληφθούν οι κρίσεις. Αυτό θα έκανε τους ε, εταίρους στην αγορά να ουσιαστικά να κάνουν ε, ε, κερδοσκοπικές πράξεις στην αγορά περιμένοντας ότι δεν θα υπάρχει ένα σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό δεν είναι θετικό. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτείας έχει βοηθήσει να αποτρέψει την, ε, την χρηματοοικονομική κατάρρευση. Αλλά Χωρί ένα τέτοιο σύστημα, το ευρώ θα είναι ανοιχτό σε κερδοσκοπικέ επιθέσει, είτε υπάρχει οικονομική βάση σε αυτέ ή όχι. Το θέμα είναι πώ θα δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό διαχείριση που αποφεύγει τι κρίσει χωρί να δημιουργεί ηθικό κίνδυνο. Αυτό δεν είναι νέο θέμα, το έχουμε αντιμετωπίσει ήδη στα πλαίσια του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Ουσιαστικά σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ισχυρέ εξαρτήσει, ισχυρέ προποθέσει ό,τι αφορά τη διαρθρωτική και δημοσιονομική πολιτική σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε δημοσιονομική υποστήριξη που δίνεται σε μια χώρα που βρίσκεται σε δυσκολία η χρηματοοικονομική αυτή υποστήριξη θα πρέπει να δίνεται μονάχα για να καλυφθούν συγκεκριμένοι στόχοι που υπελαμβάνονται στο πρόγραμμα εξυγίνηση. Δεν χρειάζεται στην Ευρώπη να εφεύγουμε και πάλι τον τροχό. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την εμπειρία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και η ιστορία δείχνει ότι οι χώρε πολλέ φορέ δεν θέλουν να πάρουν υποστήριξη από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, γιατί υπάρχουν ισχυρέ προποθέσει, έντονε προποθέσει για κάτι τέτοιο. Οι πρώτε Ευρωπαϊκέ Κεντρικέ Τράπεζε πήγαν προ αυτήν την κατεύθυνση και έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων, ενώ συγχρόνω αποτρέπει κερδοσκοπικέ επιθέσει εναντίον του συστήματο. Ο μηχανισμό διαχείριση τη κρίσεω δημιουργεί και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πιο πολύπλοκο και απαιτεί κάποιον αναλογισμό. Το θέμα αυτό είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην επίλυση των κρίσεων. Αυτό σημαίνει είναι ότι τα δημόσια χρήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διασωθούν οι ιδιωτικοί φορείς που έχουν λάβει λανθασμένες αποφάσεις. Αυτό θα συνέβαινε εάν τα χρήματα που χρησιμοποιούνται από το μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσης χρησιμοποιούνται για να αποζημιώσουν τον ιδιωτικό τομέα για τις απώλειές του και με τον τρόπο αυτό να άρουν κάθε μορφή κινδύνου. Το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά από την κρίση τη Ασία τη αποανατολή έδειξαν συζητήσει ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίο θα κάνει υποχρεωτική την αναδιάθρωση. Για ένα απλό λόγο. Η φερεγγιότητα ενό κράτου είναι μια διαφορετική έννοια από τη φερεγγιότητα μιας εταιρείας ενό χρηματοπιστωτικού ιδρύματο. Βασικά εξαρτάται από την οικονομική και πολιτική βιωσιμότητα της επίτευξης ενός πρωτογενούς πλεονάσματος του προπολογισμού ώστε να μπορέσει να σταθροποιήσει το χρέος της χώρας αυτής. Αν μια χώρα είναι δεσμευμένη σε ένα πρόγραμμα ανά, ανάκαμψης το οποίο δικαιολογεί την υποστήριξη των άλλων εταίρων της, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αφαιρέγγια και δεν μπορεί να ξεπληρώσει τα χρέη της. Για αυτή αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να χωρίσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της. Ενώ από την άλλη μεριά, αν η αναδιάρθρωση του χρέους γίνει πάρα πολύ εύκολη, τότε μπορεί αυτό να παροτρύνει τις δυνάμεις της αγοράς να κερδοσκοπούν επί του ενδεχόμενου μια τέτοια αναδιάρθρωση και επομένω να κινούνται κερδοσκοπικά εναντίον μια χώρα. Επομένω, ένα μηχανισμό αναδιάρθρωση που είναι πολύ απλό θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε μεγαλύτερο ηθικό κίνδυνο. Και η μορφή των αγορών σημαίνει ότι θα υπάρξει μετάδοση των κρίσεων σε άλλε χώρε, γιατί οι δυνάμει τη αγορά, οι εταίροι τη αγορά θα θα προσπαθούσαν να διακρίνουν ποιε χώρε κινδυνεύουν να έχουν την ανάγκη αναδιάρθρωση. Ακολουθώντα λοιπόν το, ένα έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην σημερινή οικονομία που είναι ε, ιδιαίτερα εξελιγμένη είναι άχρηστη, ε, μη επιθυμητή και ε, απίθανη η ανάγκη της αναδιάρθρωσης. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος να συμμετάσχει ο ιδιωτικός τομέας είναι να εξασφαλίσουμε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίε θα μπορέσει να έχει ένα ε, αξιόπιστο μηχανισμό ε, προσαρμογής που πείθει τις αγορές να ξαναεπενδύσουν τη χώρα αυτή. Η εμπειρία δείχνει ότι τέτοια προγράμματα που είναι επιτυχή όταν πράγματι οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί είναι επιτυχείς έχουν οδηγήσει σε ανάκαμψη της εμπιστοσύνης της αγοράς στη χώρα αυτή. Μπορεί να χρειαστεί χρόνο και μπορεί να χρειαστεί αναδιάταξη τη οικονομική υποστήριξη προ τι χώρε αυτέ, αλλά στο τέλο υπήρξε και πάλι πρόσβαση στι αγορέ. Αν λοιπόν υπάρξει μια μορφή αναδιάρθρωση ή τροποποίηση μορφή του χρέου για να υπάρξει μια βιωσιμότητα του χρέου, αυτό μπορεί να γίνει μονάχα μέσω μια συμφωνία μεταξύ πιστωτών και χρεωστών. Άλλε μορφέ δράση από τη μία ή την άλλη πλευρά θα οδηγήσουν σε νομικέ διαμάχε και μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχέ των χρηματαγορών. Από αυτή την άποψη, οι, οι ρήτρε συλλογική δράσεω από τα μέλη της, χώρης, της ζώνης του ευρώ θα διευκολύνουν τους πιστωτές και τους χρεώστες να συμφωνήσουν για την καταλμή του άκου. Αυτό ήταν και το συμπέρασμα των συζητήσεων στα πλαίσια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και είναι κάτι που μπορούμε να διερευνήσουμε και πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας άλλος τρόπος να εμπιωδήσουμε ότι οι φορείς της αγοράς ε, διασώζονται είναι να χρησιμοποιήσουμε τους ε, πόρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τον επίσημο μηχανισμό να αγοραστεί χρέος στην δευτερεύουσα αγορά και με έκπτωση όπως υπάρχει στην αγορά και όχι απλώς να υπάρξει επιστροφή του χρέους σε ονομαστική αξία. Αυτό σημαίνει ότι δεχόμαστε το λεγόμενο κούρεμα, το haircut. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία περιλαμβάνεται στι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να κλείσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινό τη δικαίου στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη και όπω λέμε στα λατινικά, pacta sunt servanda. Θα πρέπει να τηρούνται οι συμφωνίε. Και αυτό αφορά όλα τα θέματα από τη δημοσιονομική ε, πειθαρχία μέχρι την υποχρέωση των κρατών μελών να αποπληρώσουν το χρέο του. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν εξετάζουμε εξαιρέσει σε αυτέ τι αρχέ και του κανόνε, όπω παραδείγματο χάρη δυνατότητα οι χώρε να τροποποιήσουν μονομερό την αξία των, χρέο, των χρεωστικών του συμβολέων. Το ευρώ και η θεσμική του οικοδόμηση είναι ένα θέμα που περιλαμβάνει το σεβασμό του δικαίου. Οποιασδήποτε αλλαγέ θα πρέπει να ενισχύσουν αυτή την αρχή και όχι να δημιουργήσουν εξαιρέσει, Ενδεχομένω επικίνδυνε εξαιρεσει που μπορούν να υποσκάψουν τη σταθερότητα και τη συνοχή όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα um, Σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη πολλοί άρχισαν να ζητούν το λόγο για να υποβάλουν ερωτήσεις. Ε, τις ακούσουμε αφού θα έχουμε ακούσει και τον ε, Επίτροπο. Ξέρω ότι ο Επίτροπος θα έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών. Θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ θερμά για το μέγα επίτευγμα της υιοθέτηση του τελικού πλαισίου εποπτείας και για την έναρξη θέση σε ισχύ του, σε ισχύ του συγκεκριμένου προγράμματος καθώς και για αυτή την πολύ επίκαιρη ακρόαση για την οικονομική διακυβέρνηση. Το νέο αυτό εποπτικό πλαίσιο και η ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση θα συστήσουν ένα νέο, σύστημα και μια νέα τάξη οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, επιτέλους στην βάση κανόνων μιας ε, ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Και ακόμα πολλά βέβαια πρέπει να γίνουν, ακόμα και αν είναι τόσο σημαντικά τα όσα ήδη έγιναν. Να τονίσω καταρχήν την ε, οικονομική εικόνα που δίνει σε αυτή την εβδομάδα η Κομισιόν. Το βασικό μας συμπέρασμα είναι ότι η, ευρωπαϊκή, η ανάκαμψη της Ευρώπης έχει τώρα φτάσει σε μια καλή φάση, έχει γίνει πιο στεναρή και αυτάρκης σε σχέση με τις ε, Τέρες βέβαια εξαγωγές και η εγχώρια ζήτηση έχει αυξηθεί και έχει φτάσει στο 1,8% για φέτος. Η ανεργία έχει σταθεροποιηθεί και η απασχόληση επίσης αρχίζει να ανακάμπτει στα περισσότερα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα έχουμε ε, πιο στέρεο έδαφος κάτω από τα πόδια μας, αλλά φυσικά δεν υπάρχει χώρος για αυτά ρέσκια. Και αυτό κυρίως για δύο λόγους. Καταρχήν, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές ε, ε, μεγέθυνσης είναι αβέβαιες. Η μεγέθυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει, ε, έχει αργούς ρυθμούς και Επίσης το ίδιο γίνεται και με την αγορά των δευτερευόντων ε, προϊόντων εδώ στην ε, Ευρώπη. Το δυναμικό της μεγέθυνσης της Ευρώπης παραμένει σε πολύ μέτρια επίπεδα όταν είναι κάτω από το μισό της εκατό στην επόμενη δεκαετία, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό και ούτε για την Ευρώπη, ούτε για την απασχόληση, ούτε για την ευημερία είναι σαφές για όλους μας ότι δεν έχουμε ακόμα ξεμπλέξει δεν έχουμε ακόμα ξεπεράσει τις δυσκολίες και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι απαραίτητη. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης χρειάζεται πολλή δουλειά σε όλα τα μέτωπα. Ίσως θυμάστε ότι όταν παρουσίασε τις πολιτικές μου προτεραιότητες εδώ ενώπιόν σας τον Ιανουάριο ζήτησα την ενίσχυση της του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την παγίωση της δημόσιας οικονομίας και τη διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, επιπλέον ε, είπα ότι θα κάνω περισσότερη οικονομική ε, εποπτεία τόσο χρηματοοικονομική όσο και διαρθρωτική και υποσχέθηκα ότι η Κομισιόν θα επέβαλε νομοθετικές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, εννέα μήνες αργότερα, Το πιο σημαντικό είναι αυτό που εξήγησε ο Λορέντζο πολύ καλά, ότι δηλαδή χρειάστηκε να λάβουμε μέτρα άνευ προηγουμένου για να σταθεροποιήσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη και άρα λοιπόν και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνδυασμός ε, αποφασιστικής δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βοήθησε στο να περιοριστεί προκύπτουν οι διαταραχές στις ε, αγορές. Σήμερα είναι η δεύτερη επέτειο της κατάρρευσης της Lehman Brothers στις ΗΠΑ. Δραματική υπενθύμηση του είδους της καταστροφής που μπορέσαμε να αποφύγουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ε, δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν υπήρξε περίπτωση Λέμαν εδώ στην Ευρώπη. Και αυτό επετέφθη χάρη της δημιουργίας τον Μάιο των ε, διαφόρων φραγμών, Ευρωπαϊκός ε, Μηχανισμός Σταθερότητας, ε, καθώς και το πακέτο δανεισμού για την Ελλάδα. Και αυτό χάρη και στην δημοσιονομική σταθεροποίηση και παγίωση κάναμε διάφορα stress tests και επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προέβησε αποφασιστική δράση. Ο συνδυασμός όλων αυτών των μέτρων ήταν πολύ σημαντικός για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού. Ωστόσο, παραμείναμε έτοιμοι για δράση Παράλληλα με τη διαχείριση της κρίσης και την ε, δημοσιονομική ε, διόρθωση και ανόρθωση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την δημοσιονομική διακυβέρνηση εδώ στην Ευρώπη, χρηματοπιστωτική μάλλον διακυβέρνηση εδώ στην Ευρώπη. Αυτό θα, καταρχήν θα πρέπει να γίνει μέσω της αύξηση των εξουσιών ε, εποπτείας της ίδιας της Ευρωστάτ όσον αφορά τους δημόσιους λογαριασμούς των κρατών μελών. Στρατηγικά στοιχεία για την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής τον Μάιο καθώς και στο μακροσκελές πρόγραμμα περί του Ιουνίου. Ως ε, πρώτο συγκεκριμένο προϊόν αυτής της ε, πρότασης μετά από την αύξηση των ελεκτικών αξουσιών της Eurostat, το πρώτο ευρωπαϊκό οικονομικό εξάμεινο θα εισαχθεί, από την 1η Ιανουαρίου ε, φέτος. Αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και το Συμβούλιο επί τη βάση πρωτοβουλία τη Κομισιόν τροποποίησε τον κώδικα διοντολογία ώστε να γίνει όντως αυτή, το οικονομικό εξάμεινο. Αυτή, η Κομισιόν δε 29 Σεπτεμβρίου σε δύο εβδομάδες θα αποφασίσει ε, περί ενός πακέτου προτάσεων που μετατρέπουν τις πιο επίγουσες νομοθετικές προτάσεις σε συγκεκριμένα νομοθετικά μέσα, εργαλεία. Αυτό το σύστημα συγκεντρώνει την δημοσιονομική πειθαρχία του συμφώνου τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την Ευρώπη του 2020 και τον νέο μηχανισμό που εμποδίζει τις μακροοικονομικές ε, διαφορές ή ελλείψεις ισορροπίας. Η οικονομική εποπτεία δηλαδή θα γίνεται στα κράτη-μέλη τη στιγμή που πρέπει. Και αυτό είναι απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εμεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε για κοινή πολιτική και οικονομική και δημοσιονομική πριν να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν να παίξουν πολύ κρίσιμο ρόλο εδώ. Ο κύκλος των ευρωπαϊκών ε, οικονομικών εξαμήνων ξεκινά τον Ιανουάριο με μία έρευνα για την ανάπτυξη, την οποία θα εκπονεί η Κομισιόν και η οποία θα εξετάζει τις δημοσιονομικές προκλήσεις. Η έκθεση θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσα κατά τη διάρκεια μάλλον του χειμερινού Συμβουλίου Κορυφής και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρέχει ε, στρατηγικές οριζόντιες πολιτικές γραμμές για την Ένωση, για τα όλα τα κρατημέλη, αλλά και για την Ευρωζώνη. Οι σε αυτές γραμμές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κρατημέλη στα, ε, στα, στα προγράμματα σταθερότητάς τους που θα υποβάλλονται τον Απρίλιο. Η Κομισιόν στη συνέχεια θα αξιολογεί τις πολιτικές που εκθέτουν τα κράτη-μέλη στα προγράμματά τους και Εάν αυτές δεν είναι επαρκείς, θα συστήνει στο Συμβούλιο να εκδώσει συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής το καλοκαίρι για τα συγκεκριμένα κρατημέλη. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι συστάσεις να λαμβάνονται υπόψη. Στο πλαίσιο αυτό να κάνω μια πρόταση για την ενίσχυση της επιρροής του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κατά την άποψή μου θα ήταν πολύ καλό, παραγωγικό, αν μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εξ αρχής. Δηλαδή, ταυτόχρονα με την ετήσια οικονομική διάσκεψη κορυφής. Θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια κοινοβουλευτική διάσκεψη που θα συγκεντρώνει το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια ώστε να συζητήσουν τις προκλήσεις και να και να συγκρίνουν τις ε, ε, πολιτικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Η Κομισιόν από τη δικιά της πλευρά θα μπορούσε να παρουσιάζει την ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη αυτή τη διάσκεψη ώστε να ξεκινήσει μια συζήτηση περιπολιτικής ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Κατά την άποψή μου κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την ύπαρξη ενός πραγματικά γνήσιου ευρωπαϊκού πνεύματος και μιας δημοκρατικής διάστασης στην ε, στον καθορισμό της πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζω αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση να αντιλάβετε λάβετε υπόψη σας και να την εξετάσετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δύο λόγια ακόμα για το συγκεκριμένο νομοθετικό πακέτο που, θα προτείνουμε σε δύο εβδομάδες. Στόχος των προτάσεων αυτών θα είναι είναι να δημιουργηθεί η εποπτεία, η κατάλληλη εποπτεία στους προπολογισμούς ώστε να δημιουργηθούν και με τη σειρά τους κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και για την αύξηση των θέσεων εργασίας. Αυτά όλα θα βασιστούν σε δύο κύρια χαρακτηριστικά. Καταρχήν, οι μηχανισμοί θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι όταν μιλάμε δηλαδή για τον μηχανισμό επιβολής και στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται και κίνητρα αλλά και κυρώσεις. Αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο πολύ νωρίτερα και στις αρχές της υφιστάμενης διαδικασίας περί ελλείμματος. Όχι μόνο δηλαδή το να γίνεται να, να έχει το κράτος μέλος επιλογή όταν ήδη έχει γίνει ζημιά. Αυτό δεν έχει νόημα. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να είναι πιο δεσμευτικοί από ό,τι μέχρι τώρα. Δεύτερον, η εφαρμογή αυτού του κανονισμού επιβολής δεν θα πρέπει να αφήνουν χώρο για παραθυράκια ή για χαλάρωση των κανόνων. Συγκεκριμένα, πριν να δούμε την υιοθέτηση οποιασδήποτε διαδικασία, οι προτάσεις ε, για τις επιτροπές για την εφαρμογή των, του μηχανισμού επιβολή σε, σε συνδυασμό με τα διάφορα βήματα για την εποπτεία του ελλείμματο θα πρέπει να υιοθετηθούν εκτός και αν το Συμβούλιο τα απορρίψει όλα αυτά. Ε, αυτό εννοεί όταν λέει ο Λορέντζο για την ε, αντιστροφή της ε, από, του βάρους απόδειξης. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να υιοθετήσουμε τις συστάσεις της Κομισιόν, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα βέτο της ειδική πλειοψηφίας για να αντιστραφεί η συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο σημερινό πλαίσιο της συνθήκης και μπορεί να γίνει γρήγορα για τα κράτη της Ευρωζώνης επί τη βάση του άρθρου 136 ενώ και οι 27 μπορούν να προχωρήσουν σε σχέση με τη δαπάνε του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού πλαισίου και των νέων κανονισμών που σχετίζονται με το εν λόγω πλαίσιο. για να απλοποιήσουμε αυτοί οι αυστηροί κανόνες δεν θα πρέπει να είναι πιο περίπλοκοι από ότι οι κανόνες σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Οι παίκτες δεν μπορούν να αρχίσουν να συζητάνε δηλαδή τους κανόνες του παιχνιδιού με τον διαιτητή κάθε φορά που διαπράττουν σφάλμα Έχω υπάρξει παίκτη και έχω υπάρξει και διαιτητή. Και ξέρω πόσο εκνευριστικό είναι όταν αρχίζουν οι παίκτε να αμφισβητούν του κανόνε στη μέση ενό παιχνιδιού. Οι κυρώσει λοιπόν θα πρέπει να είναι μια, ε, μια αυτόματη συνέπεια. Όταν οι χώρες ε, παραβιάζουν τους κανόνες και το βάζουν σε κίνδυνο τους Ευρωπαίους εταίρους τους, θα πρέπει να είναι αυτόματη η κύρωση. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, να ολοκληρώσω με κάποιες σκέψεις για το πώς βλέπω εγώ τα επόμενα βήματα αυτής της διαδικασίας. Ε, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Ο χρόνος τρέχει. Πρέπει να προβλέψουμε μέσα για καλύτερη οικονομική διαχείριση. Αυτά να γίνουν πραγματικά και λειτουργικά όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου και αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει βέβαια και τις μικροοικονομικές ε, ανισορροπίες και το χειρισμό αυτών για τις οποίες προτείνουμε δομημένο μηχανισμό που θα εντοπίζει και θα χειρίζεται τις λήψεις ισορροπίας με προληπτικό τρόπο έτσι ώστε αν η φορολογική πειθαρχία, η λιτότητα που επιβάλλεται, η δημοσιονομική λιτότητα που επιβάλλεται σε περιπτώσεις όπως η ελληνική, αυτό θα γίνει για να προληφθούν τέτοιες ε, περιπτώσεις όπως η Ισπανία ή η Ιρλανδία που ε, υποφέρουν από μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες. Εμείς προτείνουμε και ένα πίνακα βαθμολογίας για τους οικονομικούς χρηματοπιστωτικούς δείκτες και καθώς και μια εις βάθος ανάλυση αναχώρα και όταν είναι δυνατόν θα είναι δυνατόν όταν είναι απαραίτητο θα είναι δυνατόν να δίνονται, να εκδίδονται συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα. Θα θυμάστε ίσως ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο πρότεινε το State of the Union την περασμένη εβδομάδα στην, στο Κοινοβούλιο καθώς και σε μια επιστολή στον πρόεδρο Μπούζεκ ότι δηλαδή οι νομοθετικές προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να αποτελέσουν μάλλον θα πρέπει να υπόκεινται στη νέα διαδικασία fast track για το Κοινοβούλιο. όσον αφορά την υιοθέτησή τους. Εγώ θα ήθελα να σας παροτρύνω να ακολουθήσετε αυτή την πορεία και να ζητήσω την στήριξή σας για την πρόταση αυτή. Οι υπηρεσίες σας ήδη παρουσίασαν υποχειρήματα υπέρ του επίγοντος χαρακτήρα αυτής της υπόθεσης ε, και για τις εκθέσεις του κυρίου Φέιου και φέρα που ε, όντως ε, και αυτές παροτρύνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Οπότε ας προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι μαζί να ε, πετύχουμε το εποπτικό πακέτο όπου είχαμε ένα χρόνο Μάλλον το επίτευγμα που καταφέραμε για έγκριση μέσα σε ένα χρόνο του, του πακέτου για την εποπτεία, εγώ σας προκαλώ αυτό να το εγκρίνουμε πριν φτάσουμε στις ε, καλοκαιρινές διακοπές του επόμενου χρόνου. Ε, νομίζω λοιπόν πως θα συμφωνήσετε μαζί μου πως αυτό θα είναι δυνατόν αν όλοι μαζί το προσπαθήσουμε. Τώρα, ας διατηρήσουμε την όθηση αυτή για την επιβολή της οικονομικής διαχείρισης. Είναι ένα θέμα συμπλήρωσης ε, της ήδη ισχυρή ε, νομισματικής Ένωση με μια γνήσια οικονομική ένωση. Και είναι πραγματικά η ώρα για να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις απόψεις για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Θα προχωρήσουμε τώρα. Έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας για ανταλλαγή απόψεων. Επτά ε, βουλευτές ε, έχουν ε, ζητήσει το λόγο. Άλλος παρακαλώ. Κύριε Χουντή, προβλέπεστε ήδη. ο Ραμόν, αν σε έχω, περιλάβει. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιορίσετε τις ερωτήσεις σας σε ένα λεπτό, γιατί τελείως δεν θα έχουμε χρόνο για τις απαντήσεις. Και θα πάρουμε τρεις ομάδες ερωτήσεων, ανά τρεις ερωτήσεις ε, θα δίνονται οι απαντήσεις, που και αυτές πρέπει να είναι σύντομες. Ο Φιλίπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτηση αφορά τους ε, δύο μιλητές και πρόκειται για τους ε, περιορισμένους δείκτες ή τα περιορισμένα κριτήρια τα οποία αναφέρεται. Τι πρέπει να προσέξουμε. Ε, δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο κατά νου ε, το χρέος και τα πλεονάσματα, θέλω να ακούσω την άποψη επ' αυτού, αλλά και δείκτες που θα καταδεικνύουν την έλλειψη βιωσιμότητας μιας οικονομίας. Δηλαδή ίσως εξάρτηση από μη ανανεώσιμες πηγές. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, τέτοιου είδους δείκτη και προς τον Ιταλό μιλητή. Να σας πω ότι εγώ σοκαρίστηκα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρενέβη στον ε, φόρο συναλλαγών, στον φόρο Τόμπιν. πρέπει να σας πω ότι με ξέπληξε αυτή η παρέμβασή της. Ε, και κάτι, μια τελευταία ερώτηση προς τον Όλι Ρεν. Εμείς ε, υποστηρίζουμε πλήρως αυτό που είπατε, το να εμπλακούν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού στις αρχές του εξαμήνου και πολύ μου άρεσε αυτό ότι θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το διάγραμμα. Ο κύριος Χουντής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ορισμένε ερωτήσει, αλλά επιτρέψτε μου κάποιο σχόλιο. Άκουσα για άλλη μια φορά τον Επίτροπο και τον εκπρόσωπο τη Κεντρικής, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μιλούν με αυτάρκεια όσο αφορά την ανάλυση τη κρίση και με ικανοποίηση για του χειρισμού. Θέλω να σα πω ότι αυτό προσβάλλει τη μνήμη μα και δεν απαντάει στα προβλήματα των πολιτών. Ή να το πω με την ορολογία την ποδοσφαιρική που αρέσει τον κύριο Ρένο, όπω άκουσα, είναι ένα φλίαρο παιχνίδι κέντρου και τα γκολ μπαίνουν σε λάθο αιστεία. Είσαστε απόντες από την κρίση και τώρα εμφανιζόσαστε ως αντίδοτο για να μην ξαναβρούμε κρίση, να μην ξαναέχουμε κρίση, τη δημοσιονομική πειθαρχία, την ενίσχυση με αυτό το στοιχείο της οικονομικής διακυβέρνησης. Κύριε Ρεν, σας ρωτώ, νομίζετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται με ποιο τρόπο θα κυβερνάτε. Κυβερνάτε αντιδημοκρατικά. Έχετε αφαιρέσει αρμοδιότητες και από τα εθνικά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα με θεσμικό τρόπο πάνε να αφαιρέσετε στοιχεία που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, με την αντιμετώπιση της ανεργίας κτλ. Αυτό το κάνετε. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πώς θα αντιμετωπιστεί η ύφεση, πώς θα αντιμετωπιστεί η ανεργία, πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αλληλεγγύης. Και μια τελευταία πλευρά γιατί δεν έχουμε και προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, νομίζω, επιτρέψτε μου να το πω, ότι και ένας πρωτοετής φοιτητής οικονομικών επιστημών γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι μια νομισματική ένωση προκειμένου να είναι βιώσιμη εκτός των άλλων πρέπει να υπάρχει να έχει και ένα μηχανισμό δανεισμού τελευταίας καταφυγής. Τελειώνω. Δεν νομίζετε ότι η απουσία ενός τέτοιου μηχανισμού οδήγησε στα κερδοσκοπικά παιχνίδια στην Ελλάδα και αλλού και σε αυτό έχετε ευθύνε και εσείς από την Κεντρική Τράπεζα με τις δηλώσεις αλλά και με την πολιτική που χαράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με το δανεισμό των ε, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ανέ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Σάρων. Κύριε Σμάκη, αναφερθήκατε στην παρέμβασή σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή σας. Αναφερθήκατε στις συνεχιζόμενες αμφιβολίες των αγορών, στην ανάγκη να μην διαχυθούν ξανά οι αμφιβολίες αυτές, όπως συνέβη με την αρχή της ελληνικής κρίσης. Εάν σας κατάλαβα καλά, απορρίψατε τη λύση της αναδιάρθρωσης του χρέους για τις υπερχρεωμένες οικονομίες και είπατε ότι ε, η καταλληλότερη επιλογή ε, θα ήταν η δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού προσαρμογής που θα πείσει τις αγορές να επενδύσουν, να επανεπενδύσουν στις χώρες με προβλήματα. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν και να ζητήσω και το σχόλιο του Επιτρόπου, του Όλοι Ρέν επ' αυτού. Ε, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι εξακολουθεί η πίεση των αγορών απέναντι στην Ελλάδα να είναι εξαιρετικά μεγάλη, παρά το γεγονός ότι έχει εδώ και αρκετούς μήνες συμφωνηθεί ένας μηχανισμός προσαρμογής απολύτως αξιόπιστος του οποίου όλα τα συμβαλώμενα μέρη η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα η ευρωπαϊκή επιτροπή το διεθνές νομισματικό ταμείο αναγνωρίζουν την ομαλή και επιτυχή ε, εφαρμογή. πώς ερμηνεύεται λοιπόν το γεγονός ότι η πίεση των αγορών συνεχίζει απαρέκκλητα και με ποιο τρόπο νομίζετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ενός, ε, μιας δύσκολης ισορροπίας αφενός εξυγένειας των οικονομικών και αφετέρου ανάπτυξη της οικονομίας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία στις διαδικασίες και στα κριτήρια θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω ότι ο Επίτροπος θα μας ενημερώσει περισσότερο πάνω σε αυτά. Η δική μου ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Εσείς τι πιστεύετε για τη δυνατότητα να συσταθεί ένα ταμείο για το ευρωπαϊκό χρέος, ένας φορέας αν θέλετε, ο οποίος ε, θα παρεμποδίζει το να υπάρχει μετάδοση της ασθένειας ε, της ε, δημοσιονομικής επιθαρχίας, δηλαδή ενός ελλείμματος. Θα μπορούσε να είναι ένα ταμείο το οποίο να λειτουργεί αυτόνομα στις αγορές και το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και από, ένα, από τον φόρο των διεθνών συναλλαγών. Εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά. Θα ακούσουμε τώρα τις ε, απαντήσεις. Θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στο Λορέντσο. Τέσσερα λεπτά έχει το καθένα. Αλλιώ δεν θα βρούμε χρόνο να τελειώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα εξετάζουμε στο πλαίσιο των διαδικασιών. Κοιτάξτε, στο δικό μας το έγγραφο αναφέρουμε τα κριτήρια τα οποία πρέπει να εξετάζονται τόσο από δημοσιονομική όσο και από μακροοικονομική σκοπιά να μειωθεί το χρέος, το συνολικό χρέος μιας χώρας Αυτό το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα στατιστικά δεδομένα και μεγαλύτερη βούληση για πράξη. Όσον αφορά την ε, διεθνή εποπτεία, αυτό που δεν κάναμε τελευταία χρόνια είναι να εξετάζουμε την ανταγωνιστικότητα των κρατών. Δηλαδή, ε, χώρες παρουσίασαν ανάπτυξη λόγω των μισθών, ε, λόγω διαφόρων άλλων παραγόντων, που τελικά όμως αποδείχθηκαν ότι ήταν ασταθείς αυτά πρέπει να βρεθούν στο κέντρο της μακροοικονομικής εποπτείας. Και έτσι, αν μια χώρα φτάσει σε έλλειψη ισορροπίας, υπερβολική έλλειψη ισορροπίας, ανάβει ένα λαμπάκι αν θέλετε, ένας ε, φωτεινός σηματοδότης. Και οι χώρες αυτές να αναγκαστούν να περνάνε μέσα από αυστηρή πειθαρχία για να επαναφέρουν την ισορροπία. Όσον αφορά την ερώτηση ε, για το φόρο συναλλαγών, ε, εσείς τώρα μου λέτε να σας πω τι πιστεύω για αυτό το φόρο συναλλαγών. Εγώ δεν τοποθετήκα ακόμα επ' αυτού. Όσον αφορά την άλλη ερώτηση, το ρόλο του μηχανισμού ε, καταφυγής, δανεισμού καταφυγής. Αν δείτε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τους τελευταίο καιρό, ε, θα δι, βλέπατε, θα διαπιστώνατε ότι έχουμε τεράστια προβλήματα όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση κρατών που δεν είχαν πρόσβαση στις αγορές. Και το πρόβλημα είναι ότι σε αυτές τις χώρες, σε κάποιες από αυτές, το πρόβλημα προέκυψε από λάθος δημοσιονομική πολιτική. Δημοσιονομικό είναι το πρόβλημα, όχι νομισματικής φύσεως και πρώτα απ' όλα πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα οι νομισματικές πολιτικές δεν μπορούν να λύσουν ένα δημοσιονομικό πρόβλημα. Και αν μια χώρα έχει χρεωθεί τόσο πολύ που δεν την εμπιστεύονται οι αγορές, όχι μόνο οι αγορές αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες της χώρας, τότε η ίδια η χώρα πρέπει να διορθώσει το φαινόμενο αυτό και όχι οι νομισματικές αρχές που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη χώρα. Τώρα πάμε στο τι συμβαίνει με την Ελλάδα. Κοιτάξτε, Όπω έδειξε και η εμπειρία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, χρειάζεται χρόνο. Οι αγορέ έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του προ την αγορά και οι αγορέ θέλουν να δουν μια νέα ατραπό, σωστή αυτή η ατραπό και εμεί τη στηρίζουμε. Αυτή η ατραπός θα πρέπει να στηρίζεται μήνα προ μήνα. Η πρώτη έκθεση του Διεθνού Ταμείου έκρινε την πορεία επιτυχημένη, θα εκταμιευθεί η δεύτερη δόση και πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η πορεία. Κοίταξε, ο χρόνο, η εμπειρία μάλλον έδειξε ότι χρειάζεται χρόνο με 12 μήνες ε, μέχρι να επανέλθουν αγορές. Και οι αγορές τα ψάχνουν όλα. Ψάχνουν ε, τη βούληση της κυβέρνησης που στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ε, πραγματικά μας εντυπωσιάζει αλλά και την συνέπεια στο να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Νομίζω αυτά μπορεί να πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που στηρίζει το πρόγραμμα. Λέει ακολουθήστε, συνεχίστε αυτή την κατεύθυνση και στο τέλος του δρόμου θα επανέλθουν οι αγορές. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση του φορέα ή του ταμείου για το χρέος, το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει. Και εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε αρκετά χρήματα από το φόρο διεθνών συναλλαγών. Ανεξάρτητα από το ότι ένα τέτοιο φόρο ε, θα μπορούσε να επιφέρει και μεγάλη αναταραχή για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε χρέος. Πέρα από αυτό θα υπήρχε και πρόβλημα επιμερισμού. Ποιο θα πλήρωνε τι. Ορισμένε χώρε είναι πιο πλούσιε από άλλε. Και σε τελική ανάλυση ε, θίγονται θέματα τα οποία δεν έχουμε εξετάσει. Και ε, θίγονται πολύ σημαντικά προβλήματα. Εμείς ε, κατά το παρελθόν ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουμε πει ότι αυτός ο φόρος ε, διεθνών συναλλαγών δεν είναι ο καλύτερος. Καλύτερα να φορολογούνται οι εταιρείε με βάση τα κέρδη τους και όχι με βάση τις συναλλαγές. Αυτό είναι καλύτερο. Και επιτρέψτε μου να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Στρέφομαι στον Επίτροπο. Έχουμε λοιπόν ήδη σαν σχέδιο το να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στη συνάντησή μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια του χρόνου. Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε τώρα είναι αν είναι σωστή η χρονική στιγμή αυτής της ε, συνάντησης. Ίσως πριν να την προτάξουμε λιγάκι. Μπορεί κάποιοι να πανικοβληθούν και να αλλάξουν την ατζέντα τους, αλλά κατά άλλα ίσως θα είναι καλύτερο. Ο κ. Επιτροπός, ευχαριστώ. Αν χρειάζεται αίθουσα, μπορώ να σας δώσω μια αίθουσα στην Κομισιόν για να συναντηθείτε αν δεν βρείτε τίποτα στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη διαθεσιμότητα που έχετε δείξει να αντιμετωπίσετε την ε, πρόκληση αυτή της ταχείας οδού σε σχέση με την έγκριση αυτών των νομοθετημάτων. Και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε τους στόχους που είναι πολύ σημαντικοί. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Λάμπερτ και στον κύριο Χούντης από κοινού, γιατί και οι δύο, τον κύριο Χούντι, από κοινού, γιατί και οι δύο αναφέρθηκαν στο ίδιο θέμα. Ο κύριο Λάμπερτ αναφέρθηκε στον περιορισμένο αριθμό δικτών σε ό,τι αφορά τις ε, μακροοικονομικές ανισορροπίε και τα θέματα εποπτείας. Η δική μου φιλοσοφία εδώ είναι ότι η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία και τη διόρθωση. Γι' αυτό το λόγο Χρειαζόμαστε ένα ευρύτερο αριθμό ενδεικτών και όχι μονάχα δημοσιονομικού χαρακτήρα δείκτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε 6 έως 8 ε, κομβικούς δείκτες σε αυτό το πλαίσιο, οι οποίοι πρέπει να είναι απλοί και ευλήπτοι και εύκολοι να αναλυθούν ώστε να καταδείξουν ποιε είναι οι τάσει στην οικονομική μεγέθυνση, το ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών, την, τον πληθωρισμό, το μοναδίο κόστο εργασία, την παραγωγικότητα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να καταδείξουν ενδεχόμενες ελλείψει ισορροπία σε μακροοικονομικό επίπεδο. Αλλά υπογραμμίζω ότι αυτό θα είναι μονάχα ένα τμήμα τη οικονομική εποπτεία την οποία θέλουμε να ασκήσουμε. Υπάρχουν και ευρύτερα θέματα όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση, η βιωσιμότητα σε επίπεδο περιβάλλοντος, όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 που ακριβώς στοχεύει σε κάτι τέτοιο. Για την κυρία Ποδηματά. Αναφερθήκατε στις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες στις χρηματαγορές σε ό,τι αφορά ιδίως το κρατικό χρέος της Ελλάδος και άλλων χωρών. Για τις, ε, το ερώτημα αυτό απήντησε εν μέρει ο Λορέντζο. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι χρειάζεται χρόνος για να επανέλθει και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των αγορών μετά από μια κρίση. Το ουσιαστικό όμως του κεφαλαιόδες είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται τώρα στη σωστή πορεία. Η Ελλάδα έχει επιτύχει τουλάχιστον για εφέτος εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εδραίωση των δημοσιονομικών της και έχει ξεκινήσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων δομικού χαρακτήρα μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και η μεταρρυθμίση των συντάξεων και επίσης η μεταρρυθμίση της αγοράς εργασίας. Όλα αυτά είναι απόλυτα σε ευθυγράμμιση με το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα θυμόσαστε ότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έναντι της ελληνικής κυβέρνησης είχε αρχικό σχεδιασμό τριών ετών, διάρκειας τριών ετών από το Μάιο του 2010 στο Μάιο του 2013. Βέβαια, είναι απαραίτητο και ζωτικό η Ελλάδα να μπορέσει να διατηρήσει την ισχυρή προσπάθεια μεταρρυθμίσεων τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο όσο και σε δομικό επίπεδο ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει την οικονομική της ανταγωνιστικότητα και να ξεπεράσει την τωρινή ε, αρνητική δυναμική. Ο κ. Ντομανέτσι αναφέρθηκε στην ε, επιλογή του να υπάρχει ένας φορέας για την διαχείριση του χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένως την, αυτό που παραπέμπει στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και τις ε, προσωρινές ε, συμφωνίες που ισχύουν όπως είναι το ελληνικό πακέτο για τα επόμενα τρία χρόνια και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ο οποίος έχει αυτό το χαρακτήρα τρία χρόνια το, το μάξιμο. Για μένα η καλύτερη μέθοδος που μπορεί να ακολουθηθεί είναι πρώτα απ' όλα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, πώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι μηχανισμοί και παράλληλα μπορούμε να αρχίσουμε την αξιολόγηση αυτών των οικονομικών και χρηματοοικονομικών διασφαλίσεων, ώστε να έχουμε μια καλύτερη αξιολόγηση. παραδείγματος χάρη το επόμενο έτος, το 2011, και επί τη βάση αυτής της εμπειρικής ανάλυσης σε βάθος που μπορεί να γίνει και τη εμπειρία που θα έχει εκτιθεί, μπορούμε να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη πρόταση για ένα μόνιμο μηχανισμό που θα αντιμετωπίζει και θα επιλύει τις κρίσεις. Κατά την άποψή μου, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα τέτοιο μηχανισμό καλύτερα να είναι κανείς ασφαλής και υπερβολικός ίσως από το να μετανιώνει εκ των υστέρων. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθεί και ηθικός κίνδυνος με αυτό το μηχανισμό. Ευχαριστώ πολύ, λέγει Πρόεδρος, ώστε όλοι να μπορέσουν να ε, έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν μια απάντηση. Θα επανέλθω στους έξι επόμενους ομιλητές πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές. Είναι μακρός κατάλογος, αλλά Ford, Η Βίκη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Είναι πάρα πολύ σαφές από αυτά τα οποία ελέγχθηκαν ότι χώρες όπως η Ιρλανδία είναι ακόμα μακριά από το να λύσουν τα προβλήματά τους, τα οικονομικά. Θέλω να σταθώ σε δύο θέματα. Καταρχήν το πώς ξεπερνούμε τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες όταν δεν έχει κάνει έλεγχο πάνω στην πολιτική επιτοκίων του νομισματός του και εδώ τίθεται το θέμα του αν μπορεί μια εθνική τράπεζα να έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις κεφαλοχικές ε, απαιτήσει για τις εθνικές τράπεζες και να ελέγξει έτσι την νομισματική μάζα. Αυτό προσπάθησε να κάνει η Ισπανία και δεν λειτουργήσε. Επί τη βάση λοιπόν της εμπειρίας που έχετε, είναι χρήσιμο αυτό ή όχι. Και αυτό φυσικά είναι ένα εργαλείο όταν κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τα επιτόκια του σε εθνικό επίπεδο. Ένα άλλο θέμα το οποίο τίθεται και πολλοί βουλευτές σε άλλες επιτροπές έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την έννοια των ευρωομολόγων. Και είναι σαν να πιστεύουν ότι θα φυτρώσουν από μόνα τους τα λεφτά. Εάν υπάρχει όμως ε, κάτι τέτοιο ευρωομόλογα θα πρέπει να υπάρχει κεντρική εγγύηση για αυτά. Αλλιώς χρειάζεται μια νέα συνθήκη. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί θα έπρεπε να αφήσετε να υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, ε, να υπάρχει αθέτηση πληρωμής ομολόγων μόνο και μόνο επειδή μια χώρα δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επανέλθουμε και να εξηγήσουμε γιατί ορισμένε χώρε χρειάστηκε να περάσουν σε προγράμματα λιτότητο. Αλλά είδαμε ότι στο τέλο αυτού του έτου και στην αρχή του επόμενου χρόνου πολλέ χώρε όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλανδία, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλε χώρε και η Γερμανία εξάλλου, ήδη συγχρόνω και παράλληλα ξεκινούν μια σειρά από προγράμματα αυστη... ε, λιτότητο σε δημοσιονομικό επίπεδο. Μήπω αυτό θα πρέπει να μα οδηγήσει σε ανησυχίε ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει πάντα να υπάρχει μια κεντρική τράπεζα η οποία θα σταθεροποιήσει την οικονομία. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου Υπάρχει αδυναμία στις οικονομίες μας και τα επιτόκια βρισκόνται πολύ κοντά στο μηδέν. Δεν υπάρχει πολλής χώρος ελιγμών για μια κεντρική τράπεζα να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτών των προγραμμάτων λιτότητος. θα ήθελα να αναφερθώ στον Επίτροπο κύριο Όλιρεν. Πρέπει να ομολογήσω ότι συμφωνώ με την ιδέα κάποια συνεργασίας και συντονισμού στο πρώτο αυτό ευρωπαϊκό εξάμεινο, αλλά έχω και κάποιες αμφιβολίες για το καθεστώς των κυρώσεων. Τι ακριβώς κάνει το προσωπικό της Κομισιόν σε σχέση με την επεξεργασία αυτών των κυρώσεων. Τα προβλήματα είναι και η ανάπτυξη και η απασχόληση και η απόκληση των οικονομιών και οι κυρώσεις δεν αντιμετωπίζουν κάποια από αυτά τα προβλήματα, δεν επιτρέπουν στις χώρες να συμμορφωθούν προς τις ανάγκες, Δηλαδή αν δεν συμμορφώνται προς τους στόχους οι χώρες αυτές είναι γιατί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει συμμόρφωση όταν υπάρχει απόκληση μεταξύ των οικονομιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω πρόβλημα με την νομική βάση, έχω πρόβλημα με το να κόβονται τα διαρθωτικά ταμεία για ορισμένε χώρε, κάτι το οποίο θα επηρεάσει άλλε χώρε περισσότερο από κάποιε άλλε. Και επίση με την ιδέα τη αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου, που είναι κυρώσει για τι οποίε δεν υπάρχει νομική βάση πάνω στην οποία να λειτουργήσει η Κομισιόν. Και έχουμε επίση και κυρώσει οι οποίε δεν θα εφαρμόζονται ποτέ σε μεγάλε χώρε. Αυτό επομένως ίσως θα θέσει σε μεγάλη δυσκολία και θα μειώσει την αξιοπιστία της Κομισιόν και όλου του προγράμματος. Γιατί λοιπόν δεν γίνονται προσπάθειες για ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, για ευρώ ομόλογα και για μια στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης που χρειαζόμαστε, τον Διόγκο. Ευχαριστώ, θα ήθελα να ξεκινήσω Ευχαριστώ τους ομιλητές. Και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για τα λόγια που είπε σε σχέση με την έκθεση που συζητείται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, που είναι μια έκθεση που έχει συνταχθεί με την προσπάθεια όλων των πολιτικών ομάδων και με στόχο το Κοινοβούλιο να αποκτήσει μια ξεκάθαρη φωνή σε σχέση με αυτό το θέμα. Κύριε Επίτροπε, το πρώτο σύνολο ερωτήσεων που εγώ ήθελα να υποβάλω έχει να κάνει με το θέμα των κυρώσεων. Και θέλω να καταλάβω αν σε αυτές οι κυρώσεις που προτείνετε είναι κυρώσεις όπως αυτές που προβλέπονται αυτή τη στιγμή από τη συνθήκη, αν ε, θεωρείτε πως η σε σχέση με αυτό το θέμα ε, θα γίνει νέα νομοθεσία ή αν αυτό ε, θα αφορά περισσότερο πολιτικής φύσης κυρώσεις ή οικονομικής φύσης κυρώσεις που θα σχετίζονται με τους σπόρους. Σε δεύτερο επίπεδο, σε επίπεδο εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αυτό που διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι είχε μεγάλη σημασία για το κριτήριο της, του ελλείμματος, ενώ έχει ξεχαστεί το κριτήριο του χρέους. Πώς βλέπει ο Επίτροπος το ζήτημα μιας ειδικής, ε, ε, μάλλον μιας μεγαλύτερη σημασία που θα δοθεί στο θέμα των, του χρέους. Και τώρα, σε σχέση με την διακυβέρνηση την οικονομική έκθεση ΣΤΑΕΣ που έχει στόχο να ε, δούμε με βάση τη συνθήκη αν αυτό είναι θέμα μέσο ή προθεσμο Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φέιο είναι συγητής για την έκθεσή μας για αυτό το θέμα. Ο Σβέν. Καταρχήν στον κύριο Μπενισμάγκη να διευκρινίσω η δική μου παρατήρηση αφορούσε τις ε, πολύ έντονες δηλώσεις του Προέδρου σας τελευταίο ΕΚΟΦΗΝ που έλαβε πολύ σταθερή θέση σε σχέση με τον ε, φόρο δημοσιονομικών ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για να επανέλθω στο ερώτημα του συναδέλφου για τα όσα είπε ο Όλη απόλυτα τα συμμερίζομαι θα πρέπει να δούμε τους αριθμούς ε, στις οικονομικές αγορές πρέπει να ενεργήσουμε ε, γρήγορα ε, αν θέλουμε να βρούμε ένα νέο καθεστώς για τη διεύρυνση της του καθεστώτος της οικονομικής διακυβέρνησης. Για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για κάτι τουλάχιστον για μένα, Υπάρχουν δύο βασικές γραμμές ε, ε, ερωτήσεων. Δηλαδή, πώς θα μοιραστεί το φόρτος όταν ε, υπάρχουν ανισορροπίες και αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια συνένεση πως ο φόρτος θα βαρύνει αυτούς που έχουν ελλείμματα. Αυτό είναι ένα θέμα κλειδί. Πώς θα βοηθήσουμε τις χώρες που είναι πολύ χρεωμένες να, να αποπληρώσουν το χρέος τους με ε, επιτόκια που τα οποία να είναι προσιτά και έπειτα ποιος ε, θα εξισορροπήσει τους εμπορικούς ε, λογαριασμούς, τα ισοζύγια. Αυτό σημαίνει πως ε, δεν θα μπορεί να γίνει αυτό με τις χώρες που έχουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει να γίνει και μια συμβολή από μεγαλύτερη ζήτηση, μέσω μάλλον μεγαλύτερη ζήτηση από τις άλλες χώρες. Παρακαλώ, μην βλέπετε μόνο τη γη προς τη Γερμανία. Ε, κοιτάξτε το κοινό συμφέρον της Ευρώπης γιατί διαφορετικά θα έχουμε τεράστιες δυσκολίες για να βρούμε συνένεση και να έχουμε μια, ένα νέο σύστημα διακυβέρνηση για την Ευρώπη. Θα μπορούσα να τα έχει πει πιο σύντομα, αγαπητέ. Ωραία, μόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση για τον ε, εκπρόσωπο της ε, ΕΚΤ και τον Επίτροπο. Σύμφωνα με τους ε, στατιστικές της Τράπεζας της Ισπανίας, το, οι πιστώσεις των τραπεζών μειώνονται το 2010. Χωρίς να ξεκινήσει μια ε, ροή πιστώσεων, θα υπάρξει οικονομική ανάκαμψη. Κατά τη γνώμη μου, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει η Ισπανική κυβέρνηση γίνονται χωρίς αρκετή πεποίθηση. Στο όνομα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης ίσως να χρειάζεται περισσότερο παρεμβατισμός στην Ισπανία που θα προέρχεται όμως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς το πιστεύετε αυτό ή όχι. Σας ευχαριστώ. Θα, θα δώσω πρώτο το λόγο στο Λορέντζο γιατί ξέρω ότι πρέπει να φύγει. Έχει το λόγο. Εντάξει, σε 10 λεπτά πρέπει να φύγω, οπότε μπορώ να απαντήσω για το θέμα του πώς μπορεί κανείς να λύσει τις μακροανισορροπίες αν δεν μπορείς να σε ελέγξει τα επιτόκια. Όλες οι χώρες που μπήκαν στην Ευρωζώνη το γνωρίζουν αυτό. Οπότε πρέπει να εξοπλιστούν με εργαλεία για να το αντιμετωπίσουν το θέμα. Και αν δει κανεί την υπόθεση τη Ιρλανδία, εγώ μπορώ να σκεφτώ μια ολόκληρη σειρά μέτρων, αρχίζοντα από τη φορολογική πολιτική, που είναι πολύ θετικά και ευνοϊκά για τι κατασκευέ και για το χρέο. Ε, για ρυθμιστικά μέτρα, ώστε να καθοριστεί καλύτερα πώ πιστώνουν οι τράπεζε. Όμως ε, αυτά όλα τα έχουν απο... είναι ευθύνη των κρατών μελών. Βασίσαν ε, τα ίδια τα κρατημένα να κρατήσουν αυτές τις ευθύνες. Δεν είναι σωστό να λέμε λοιπόν πως δεν υπάρχουν μέσα εργαλεία επειδή δεν έχουμε το επιτόκια. Εντάξει, τα επιτόκια τα χειρίζεται η ΕΚΤΑ, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ανισορροπίες. Ε, λοιπόν, ε, νομίζω πως η Νομισματική Ένωση Ναι, έχει δοθεί πολλή κυριαρχία σε θέματα νομισματικά, αλλά μεγάλο τμήμα της κυριαρχίας παραμένει στα χέρια των κρατών μελών. Τώρα, αυτά που είπατε για τα ευρωομόλογα τα συμμερίζομαι. Και να πούμε τώρα για τις συναλλαγές. Αυτά που είπε ο Πρόεδρος, δηλαδή την αντιστροφή του φόρου για τις συναλλαγές. Καταρχήν αυτό που ανέφερα νωρίτερα, είναι αυτή η βάση για να χορηγηθούν να, κατανε... Μάλλον, να έχουμε έναν αποτελεσματικό φόρο. Μήπω είναι καλύτερο να φορολογηθούν τα κέρδη και όχι οι συναλλαγές. Δεύτερον, χρειάζονται τράπεζες για να, μπορούν, να, μπορεί να γίνει ε, εκ νέου κεφαλαιοποίηση και να μπορέσουν να παρέχουν πιστώσεις στις αγορές. Αν τους φορολογήσουμε και άρα τους αφαιρέσουμε πόρους, αντί αυτοί να πάνε στη νέα κεφαλαιοποίηση, αποδυναμώνονται οι τράπεζες που αντίθετα θα έπρεπε να μπορούν να ε, χρησιμοποιούν εκ νέου τα κεφάλαια. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για την επιβολή τέτοιου φόρου. Ίσως να είναι καλό ένα τέτοιο μέτρο στους ε, τους καλύτερους, αλλά όχι στη κρίση την οποία διανύουμε τώρα. Τις περισσότερες φορές λοιπόν κάτι τέτοιο θα γίνει μέσω του προϋπολογισμού. Καλύτερα είναι δηλαδή να υπάρξει ένας φόρος για να δημιουργηθεί ένα ταμείο ώστε να αποφεύγονται τέτοιες δυσκρίσεις. Για τις κυρώσεις, οι, κυρέ, οι κυρώσεις αφορούν τον όλοι, αλλά εγώ να πω ότι οι κυρώσεις δεν βοηθούν να δημιουργηθεί απασχόληση και ανάπτυξη, αλλά αυτό που βοηθούν είναι να αποφευχθούν οι πολιτικές που δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για την ε, δημιουργία τέτοιου ε, κλίματος. Δεν αρκούν, αλλά χρειάζονται, γιατί διαφορετικά υπάρχει ο πειρασμός να εφαρμοστούν πολιτικές που μετά με τη σειρά τους γίνονται φάρος για τους γείτονες και μετά αναγκάζεται να ζητήσεις βοήθεια από τους γείτονες. Καλύτερα είναι λοιπόν να προλαβαίνει κανείς παρά να προσπαθεί να μετά να ε, διορθώσει τα στραβά. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ισπανία συμβαίνει σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Είμαστε στην ίδια κατάσταση με τις πιστώσεις, είναι ακόμα αρνητικές. Έχουμε δει κάποιες πιστώσεις σε κάποιες χώρες, ιδιαίτερα στον τομέα των ε, νοικοκυριών, αλλά η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη και γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε βέβαιοι ότι οι, χώρες, οι τράπεζες συγγνώμη, να διαρθρώνονται ε, και ε, κεφαλαιοποιούν εκ νέου. Νομίζω με την ευκαιρία να πω ότι στην Ισπανία κάνουν πολύ καλή δουλειά γιατί η αναδιάρθρωση που γίνεται στην Ισπανία ε, προχωρεί προς την σωστή κατεύθυνση αλλά θα πάρει χρόνο, δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει άμεσα. Όσον αφορά τις ε, πρώτες ερωτήσεις που κάνετε σχετικά με τις ε, μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες και τα προγράμματα λιτότητας. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα των της ανεξάρτητης πολιτικής ε, επιτοκίων στο οποίο αναφερθήκατε και πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την έλλειψη ισορροπίας. Είναι γεγονός ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αποφάσισαν να επιλέξουν ε, το κοινό νόμισμα και κοινή μοίρα τόσο στα οικονομικά όσο και στα νομισματικά και τα πολιτικά θέματα που αφορούν στα κράτη-μέλη. Και βεβαίως αυτό συνεπάγεται εκούσια παρετήθηκαν της ε, κυριαρχικής τους, ε, κυρίαρχης πολιτικής τους στα επιτόκια, εκχώρησαν αυτή την αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όσο λοιπόν υπάρχει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, κυρίως ε, η Ευρωζώνη, το συμπέρασμα που προκύπτει ότι αυτό ήταν εποφελές για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Παράλληλα βέβαια, είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε ε, κάποιες ε, άλλες πολιτικές, ε, άλλους τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εμφανίζονται αρνητικές ανισορροπίες. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές άλλες πολιτικές αλλά και δείκτες που μπορούν να προσφέρουν έγκαιρη προειδοποίηση οποτεδήποτε εμφανίζονται μακροοικονομικές ανισορροπίες, φούσκα ακινήτων ή αποκλήσεις μείωση της παραγωγικότητας, αύξηση του, της ε, μονάδας κόστος εργασίας. Υπάρχουν λοιπόν αυτά, αυτές οι δυνατότητες. Όμως, επαναλαμβάνω, ήταν εκούσια η επιλογή των κρατών μελών να επιλέξουν την κοινή πολιτική. Ε, θα μπορούσαν να υπάρξουν και πολλές άλλες πολιτικές που θα επηρέαζαν ε, την ανταγωνιστικότητα και την ε, πολιτική τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα την αναφορά σας στα ευρωομόλογα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε ομόλογα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραδείγματο χάρη ο κύριος Μπαρόζο την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο, μίλησε για ομόλογα που προσφέρονται για επενδύσεις. Αυτό είναι απόλυτα θετικό και αν πραγματικά θέλουμε την οικονομική ανάπτυξη και τη θέλουμε, πρέπει να αναζητήσουμε καινοτόμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, ε, ΣΔΙΤ, συμπράξει δημόσιο-ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εξυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την απασχόληση αλλά και προγράμματα μεγάλης κλίμακας. Εχθές λοιπόν Είχαμε μια εσωτερική ομάδα εργασία ε, στην Επιτροπή. Ο κύριος Φίλιπ Μέστρατ από την ERB, ε, την Τράπεζα Ανασυγκρότηση, ε, παρουσίασε τι απόψει του. Εμεί συνεργαζόμαστε στενά με την Τράπεζα Ανασυγκρότηση και του επόμενου κάνα δύο μήνε θα καταθέσουμε συγκεκριμένε προτάσει μέχρι ε, τα τέλη Δεκεμβρίου ενώ πιο συγκεκριμένα. Δουλεύουμε πολύ ε, ουσιαστικά πάνω σε αυτές τις προτάσεις για να ε, μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο που προβλέπει, προβλέπει τα ευρωομόλογα. Όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις, κάτι που το ανέφεραν αρκετοί ομιλητές και ο κύριος Φέγιο, κατά τη δική μου άποψη είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε τόσο την ε, δημοσιονομική πειθαρχία όσο και αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις που θα ε, οθήσουν, προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Αν δούμε λοιπόν τις ε, κυρώσεις και αν δούμε τα θέματα που έθιξε ο κύριος Φέγιο που το θέμα κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει νέα νομοθεσία ή όχι, η απάντηση είναι ναι, πράγματι, νέα δευτερογενής νομοθεσία και δεν θα καταθέσουμε προτάσεις που αφορούν την αλλαγή των συνθήκων. Πρέπει να διατηρηθεί ο δυναμισμός που υπάρχει να διατηρηθεί από το σύστημα της οικονομικής διακυβέρνησης και γι' αυτό το λόγο εμείς προτιμούμε την δευτερογενή νέα και αναθεωρημένη δευτερογενή νομοθεσία για να επιτύχουμε το στόχο μας και στο πλαίσιο αυτού του νομοθετικού πακέτου θα καταθέσουμε μία πρόταση ε, γι' αυτό το, την αντιστροφή του συστήματος ε, πλειοψηφικού, ε, πλειοψηφικού συστήματος Επίσης ε, θέσετε το ερώτημα κατά πόσον θα υπάρχει μια ξεχωριστή διαδικασία αντιμετώπισης χρέους. Εμείς προτιθέμεθα να προτείνουμε ε, το στοιχείο του χρέους σε αυτό το σύμφωνο σταθερότητας που ανέκαθεν υπήρχε αλλά ποτέ ε, δεν είχε εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε, αν τελικά το Συμβούλιο εγκρίνει την πρότασή μας, είναι αυτό το κριτήριο περί χρέους πράγματι να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη σε αυτή τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Νομίζω ότι ήδη απάντησα στην ε, ερώτησή σας ε, για τις ε, αλλαγές στη συνθήκη. Η Κομισιόν επιθυμεί να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν. Αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί από τον κύριο Χέρμαν Φαρόμπαϊ. Έχω χρόνο. Δεν θα απαντήσω στον κύριο Κίκολ την άλλη φορά. Ε, να τελειώσω όμως λέγοντας, εσείς είπατε ότι υπάρχουν και κάποιοι γερμανικοί όροι που επιβάλλονται και κλεισμένων των θυρών. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Αν εσείς ξέρετε να μου το πείτε, να έρθετε να μου το πείτε. Η δική μου άποψη είναι ότι το σημαντικότερο είναι τέτοιου είδου απόκληση ανταγωνιστικότητα που έχουμε διαπιστώσει, όπω παραδείγματο χάρη στην περίπτωση τη Ελλάδα αλλά και άλλων χωρών στην Νότια Ευρώπη, είναι σημαντικό οι χώρε που έχουν και αυτέ πλεονάσματα να αναζητήσουν και αυτές διαρθρωτικές αλλαγέ για να ενισχύσουν ε, την ε, κατανάλωση τη ζήτηση τη οικονομία του. Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Οποτεδήποτε κάνουμε αναλύσεις και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας και προσβλέπω στο να συνεχιστεί η συζήτηση για το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Μερσή κύριε Επίτροπε. Συγγνώμη που σας πίεσα λιγάκι χρονικά στο τέλος. Αλλά αν είναι μακροσκελής η ερώτηση πρέπει να έχει απάντηση. Περνάμε τώρα στο, στη συζήτηση του πάνελ και με μεγάλη χαρά θα, θα καλωσορίσω όπως είπα και στην αρχή τους τρεις ομιλητές μας οι οποίοι έρχονται σιγά σιγά στο Προεδρείο. Επίσης θα καλέσω ένα από τους αντιπρόεδρους να με αντικαταστήσει γιατί πρέπει να πάω να ε, διευθύνω ένα τριγωνικό διάλογο. Μερικές φορές λοιπόν είναι χρήσιμο να προσπαθήσουμε να βρούμε σε, να φτάσουμε συμφωνία για τα πράγματα αυτά όπου μπορεί να εξεύρουμε συμφωνίες. So uh, Αναδιαθρώνουμε λοιπόν την, ε, το Προεδρείο μας. Έχουμε τον Κάρλο Κοτορέλη που είναι επικεφαλής του Τμήματος Δημοσιονομικών Θεμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Στεφάν Κολινιόν που τον ξέρετε πολύ καλά από την ε, σχολή Σαντάνα των ε, προ... προχωρημένων σπουδών και τον κύριο Σαπίρ επίσης και ο κύριος Στόιαν θα αναλάβει το Προεδρείο στην θέση εμού της Ιδίας. Ξεκινάμε αμέσω τη συζήτηση του πάνελ και θα ζητήσω και από τους τρεις που είναι τα μέλη του πάνελ να μιλήσουμε μεταξύ 10 και 15 λεπτά ώστε να επιτρέψουμε σε όλους τους συμμετέχοντες, συμμετέχοντες μάλλον, να θέσουν ερωτήσεις και να υπάρχει και χρόνος για απαντήσεις. Δίνω το λόγο στον κύριο Κάρλο Κοταρέλη που είναι ο που είναι μέλος του Δημοσιονομικού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και έχει να μας δώσει ορισμένε ιδέες για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις. Χαίρομαι κύριε Κοταρέλη που είσαστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε. Το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα είναι η βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ευρύ και δύσκολο θέμα. Υπάρχουν πολλές προτάσεις, υπάρχουν πολλές απόψεις. Θα είναι αδύνατο για μένα να μπορέσω να συνοψίσω και να σχολιάσω όλες αυτές τις απόψεις οι οποίες έχουν διατυπώθει. Γι' αυτό εγώ θα εστιάσω στο συγκεκριμένο θέμα της διακυβέρνησης στο δημοσιονομικό τομέα στην περιοχή του ευρώ. Γιατί πιστεύω ότι εδώ βρίσκεται το κέντρο της συζήτησης, μάλλον εδώ είναι πιο έντονη η συζήτηση και είναι εδώ μεγαλύτερη ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Θέλω να αντιμετωπίσω δύο βασικά θέματα. Καταρχήν, τι έχει πάει στραβά <clears throat> με το τωρινό σύστημα, με το τωρινό πλαίσιο και το δεύτερο ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ξεκινώ λοιπόν με τα προβλήματα του τρέχοντος πλαισίου για την δημοσιονομική πολιτική και διακυβέρνηση. Πρέπει καταρχήν να αναγνωρίσουμε ότι από την αρχή, αυτό ήταν γνωστό από την αρχή, ότι ήταν πολύ δύσκολο το να υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο. Πριν από 20 χρόνια ξεκίνησε η συζήτηση με την αναγνώριση δύο αναγκών. Πρώτον, το να υπάρξει επαρκή ευελιξία για τι δημοσιονομικέ πολιτικέ των μεμονωμένων χωρών, γιατί με την ε, μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση της νομισματικής πολιτικής, η δημοσιονομική πολιτική ήταν ο κύριος τρόπος με τον οποίο μπορούσε μια χώρα να αντιμετωπίσει συγκεκριμένους κλειδονισμούς. Από την άλλη πλευρά υπήρξε μια αναγνωρισμένη ανάγκη να υπάρχουν κοινά πρότυπα, κοινά και υψηλά πρότυπα για δημοσιονομική υπευθυνότητα από κάθε μεμονωμένη χώρα μέλος. Γιατί ήταν γνωστό από την αρχή ότι τα προβλήματα και η κρίση στο δημοσιονομικό τομέα σε οποιαδήποτε χώρα όσο μικρή και να είναι, θα οδηγούσε σε κλειδονισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό όλες οι χώρες είναι πολύ σημαντικές για να μπορέσουν να αποτύχουν, να τους επιτρέψουμε να αποτύχουν. Έχουμε φυσικά το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου σε αυτήν την περίπτωση και υπάρχει η ανάγκη να έχουμε κανόνες οι οποίοι θα περιορίζουν τη δημοσιονομική πολιτική για όλες τις χώρες. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα των τελευταίων μηνών έδειξαν πόσο ισχυροί μπορεί να είναι αυτοί οι που προέρχονται από μία και μόνο χώρα. Βέβαια, η κρίση της Ελλάδος δεν προεβλέπεται να συμβεί καταρχήν. Και το ερώτημα είναι τι πίεση στραβάκι. Εδώ νομίζω ότι υπάρχουν τρία κύρια κενά και τρία κύρια χάσματα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Καταρχήν, το ο λεγόμενος βραχίων πρόληψης που έχει σαν στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έχει σαν στόχο να προλάβει τα δημοσιονομικά, τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα και ανισορροπίες. Δεν λειτουργήσε, αλλά αυτό γιατί δεν υπήρχε κάποιο ε, δεσμευτικό νομικό εργαλείο που θα κρατούσε υπόλογες τις κυβερνήσεις για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων τους και για την μείωση του υπερβολικού χρέους ή ελλείμματος με ένα ικανοποιητικό τρόπο. Ως εκ τούτου δεν υπήρχαν αρκετά αποθέματα τα οποία να έχουν δημιουργηθεί σε καιρούς παχαίων αγελάδων που θα μπορούσαν να απορροφήσουν και τον αντίκτυπο της κρίσης για τα δημοσιονομικά των κρατών μελών. Ένα δεύτερο χάσμα, ένα δεύτερο κενό είναι ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που μπορούσε να υπάρχει κάποια δράση γιατί οι χώρες ξεπερούσαν το 3% σε επίπεδο δημοσίου ελλείμματος αυτή η δράση, η επιβολή του μηχανισμού αυτού για, τα υπερβολικά ελλείμματα δεν έλαβε χώρα. Υποσκάφθηκε από πολιτικές θεωρήσεις που είχαν να κάνουν με, την, το γεγονός ότι είναι το Συμβούλιο που έχει την, τον τελικό λόγο για τα θέματα αυτά και η αντιμετώπιση η αντιμετώπιση της πρόσφατης κρίσης δείχνει ακριβώς πόσο δύσκολο είναι να εφαρμοστούν οι πτυχές του μηχανισμού επιβολής κατά των ε, υπερβολικών ελλημάτων μεταξύ των οποίων των κυρώσεων και ακόμα και η μεταρρύθμιση του μηχανισμού αυτού το 2005 δεν αντιμετώπισε καθόλου το θέμα της ε, ικανότητας επιβολής. Αντίθετα, έθεσε ακόμα μεγαλύτερη ευκαμψία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των χωρών με υπερβολικό έλλειμμα. Τρίτο κενό, τρίτο πρόβλημα μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ή ήταν η απουσία μιας ικανότητας διαχείρισης των κρίσεων και επίλυσης κρίσεων, λέω ήταν γιατί με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μέσου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό το κενό αυτό. Οπότε θα εστιάσω Θα ασχοληθώ λοιπόν με το πρόβλημα της ενίσχυσης του προληπτικού βραχίωνα της εποπτείας και την, το θέμα της επιβολής κυρώσεων Αυτά τα δύο θέματα λοιπόν, η πρόληψη και η επιβολή κυρώσεων συνδέονται. Ένα από τα προβλήματα με τον ε, να πρόληψη είναι ότι δεν υπήρχαν τρόποι να εφαρμοστεί, να υπάρξει υλοποίηση αυτής της προστασίας. Ξεκινώ λοιπόν στην παρουσίασή μου με την άλλη πτυχή πρώτα, την αστυνόμευση και την επιβολή. Για να είναι αξιόπιστη η επιβολή, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Αλλά για μένα είναι το πιο σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να εδραιώσουμε την δημοσιονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάω για αστυνόμευση και επιβολή αποφάσεων, εννοώ το να μπορεί να ληφθεί μια απόφαση ότι είναι υπερβολικό το έλλειμμα μιας χώρας και να υπάρξει επιβολή κάποιας μορφής κυρώσεων ως αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης. Εδώ το κύριο ζήτημα κατά την ε, <clears throat> απόψή μου είναι το ποιο θα έπρεπε να έχει την ευθύνη του να παίρνει αυτή την απόφαση και να καταλήξει το συμπέρασμα ότι είναι υπερβολικό το έλλειμμα. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να αποφύγουμε να γίνεται πολιτικό παζάρεμα όπως αυτό έγινε μεταξύ του 2003 και του 2005 και το οποίο ουσιαστικά οδήγησε στην παράλυση του συστήματος αυτού του δημοσιονομικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο στην περίπτωση αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω και να δώσει αυξημένη αρμοδιότητα για τη λήψη αυτής της απόφασης είτε στην Κομισιόν είτε σε ένα αλεξάρτητο φορέα ο οποίος θα πρέπει να δημιουργηθεί για το φορέα αυτό. Βέβαια το Σύμβουλο μπορεί να διατηρήσει κάποιες εξουσίες ανησυχηρίας που να ε, απαιτούν είτε ομοφωνία είτε μια ενισχυμένη πλειοψηφία. Αυτός λοιπόν ο κύριος τομέας μεταρρύθμισης που είναι απαραίτητος. Υπάρχει ένας άλλος τομέας που πρέπει να λάβουμε υπόψη γιατί το τωρινό σημείο αφορά άμεσες κυρώσεις σε χώρες οι οποίες έχουν ένα έλλειμμα. <clears throat> Αυτό θα κάνει τις κυρώσεις λιγότερο πιστευτές. Μια λοιπόν ιδέα που είναι ενδιαφέρουσα είναι να υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών, δηλαδή να υπάρχουν κυρώσεις υπομορφή καθυστέρησης πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το θέμα της ε, βελτίωσης του βαρχείων απρόληψης, εγώ θα πρότεινα μία προσέγγιση τριπυλωνικού χαρακτήρα. Ο πρώτος πυλώνας θα σήμαινε να έχουμε δεσμευτικά νομικά εργαλεία για να ενθαρρύνουμε τις χώρες να έχουν ένα ευρία τιενία ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξασφαλίσει κάτι τέτοιο. Ένας τρόπος είναι να έχουμε δημοσιονομικές κυρώσεις ή δημοσιονομικά κίνητρα που να σχετίζονται με αυτό το βραχείο. Δηλαδή όλα αυτά να γίνονται πρωτού φτάσει μια χώρα το 3% σε επίπεδο ελλείμματο. Δεύτερος τρόπος είναι να ενεργοποιείται η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο. <laughs> ακόμα και πριν το έλλειμμα ξεπεράσει την τιμή αναφορά των 3%. Μια δυνατότητα η οποία είναι πιστεύω εφικτή είναι να εξετάσουμε να ξεκινούμε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος όταν το χρέος μιας χώρας ως ποσοστό του ΕΠ ξεπερνάει το 60% και δεν μειώνεται αρκετά γρήγορα. Καταρχήν, θα έπρεπε να είναι δυνατό να τροποποιήσουμε και το όριο αναφοράς του 3% με το να καθορίσουμε ως ε, έλλειμμα αναφοράς κάθε χρόνο ένα έλλειμμα που να αντιστοιχεί σε ένα διαρθωτικό, διαρθωτικά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό όπως αυτό το καθορίζουν οι υπηρεσίες της Κομισιόν. Φυσικά μια τέτοια μεταρρύθμιση της συνθήκης θα απαιτούσε ομοφωνία των κρατών μελών. Ο δεύτερος μεταρρυθμιστικός πυλώνας <clears throat> μέσα στα πλαίσια του βραχίων απρόληψης και εποπτείας είναι μια εξέλιξη που έχουμε ήδη δει να λαμβάνει η χώρα, δηλαδή να βελτιώσουμε την πρόληψη με το να διευρύνουμε την εμβέλεια των υπείων εργαλείων που έχουν να κάνουν με την εθνική οικονομική πολιτική. Αυτό νομίζω ότι είναι η βασική ιδέα πίσω από το ευρωπαϊκό εξάμεινο. <clears throat> νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό και θετικό βήμα, διότι θα επιτρέψει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς να διαδραματίσουν ένα πιο σημαντικό ρόλο σε εθνικό επίπεδο για την διαμόρφωση της ε, δημοσιονομικής πολιτικής της εθνικό επίπεδο. Τρίτος πυλώνας πρόληψης και εποπτείας θα ήταν το να βασιστούμε περισσότερο στο να παροτρύνουμε και να κάνουμε ενδεχομένω υποχρεωτική την έγκριση δημοσιονομικών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα σήμαινε ότι τα κράτη-μέλη θα νιώθουν περισσότερο δεσμευμένα από αυτούς τους κανόνες και αυτό πιστεύω ότι είναι πράγματι και μία η υποχρέωση η οποία απορρέει από το πρωτόκολλο της συνθήκης για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και θα μπορούσε με κάποια οδηγία να επεκταθεί σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη <clears throat> ε, όθηση που έχει δοθεί στην εφαρμογή τέτοιων κανόνων μετά από τις αποφάσεις που ελέγχθησαν στην Γερμανία και μετά στη Γαλλία για την εφαρμογή νέων δημοσιονομικών πλαισίων. Μία τελευταία παρούς, παρατήρηση. Έχω μιλήσει αρκετά για τις κυρώσεις και για τις ε, δεσμευτικές επιβολές περιοριστικών μέτρων Αναρωτιέμαι πως πρέπει να μιλήσουμε και για καρότα, για την εφαρμογή θετικών μέτρων τα οποία θα αμύψουν την καλή συμπεριφορά των κρατών μελών. Μία δυνατότητα προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν να δημιουργηθεί σε ε, ε, κεντρικό επίπεδο της, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μια κοινή δεξαμενή κονδυλίων ώστε οι χώρες που έχουν καλή δημοσιονομική συμπεριφορά μπορούν να αντλήσουν κονδύλια. Από εκεί, παραγωγικά, αυτό μπορεί να είναι ένα τμήμα των εσόδων <clears throat> ε, ΦΠΑ ή εσόδων από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Αυτό δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη και λεπτομεριακά, αλλά είναι μια ιδέα που αξίζει να την εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Στεφάν Κολινιόν, καθηγητή οικονομικών στο... στην σχολή Σεντάνα της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη είναι σε ένα όριμο στάδιο. Πολλές από τις προτάσεις που βρίσκονται επιτάπητος και προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κομισιόν, ε, λιγότερο από το Κοινοβούλιο αλλά και από τα κράτη-μέλη όπως η γαλλογερμανική δήλωση, φαίνεται να το θεωρούν κυρίως ως ένα τεχνικό θέμα. Συζητούν νέα μέσα, νέα εργαλεία αλλά βασικά πρόκειται για μια τεχνοκρατική, ένα τεχνοκρατικό εγχείρημα το οποίο συζητείται ανάμεσα σε γραφειοκράτες, δηλαδή πώς ε, θα ελέγχουν καλύτερα αλλήλους. Ε, βασικά χρειάζονται όλα αυτά τα εργαλεία νομίζω πως, ε, δεν έχει, πως έχει το βασικότερο ερώτημα η μόνη φορά που είχα κάποιον που μίλησε από κάποιο βασικό ε, θεσμικό όργανο ήταν αυτά που ακούσαμε μόλις από τον κύριο Κονταρέλη. Ε, είναι το θέμα του όπως το έθεσε εκείνο. η αποτυχία ήταν ότι δεν υπήρχαν δεσμευτικά εργαλεία ώστε οι κυβερνήσεις να προβούν στο έργο τους. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί μια ομάδα κρατών μελών να πει σε κάποιο κράτο μέλος τι να κάνει αν έχει εκλεγεί για να κάνει κάτι άλλο. Και αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το ερώτημα, τότε η Ευρώπη πάει ίσια σε αδιέξοδο. Πάει κατευθείαν σε αδιέξοδο. Οι δεσμευτικέ διαδικασίε είναι σημαντικέ, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν υπάρχει νομιμότητα πίσω από αυτέ. Η Ευρώπη υποφέρει από κακή απόδοση των πολιτικών. Ο Τόνι Μπλερ ήρθε μια φορά στο κοινοβούλιο και είπε ξέρουμε να κάνουμε, τι να κάνουμε και κάνουμε το σωστό. Βλέπουμε όμως ότι σωστά, οι σωστές ενέργειες δεν γίνονται οι πολιτικές ε, έχουν αποτύχει και έχουν ε, δεν έχουν σταθεί εντάξει των Ευρωπαίων πολιτικών και αυτό γιατί απαραίτητα οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε και όλα αυτά υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και υποβαθμίζουν, υπονομεύουν την συστή διακυβέρνηση των κοινών αγαθών Πράγμα που όλοι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί επιθυμούν, ε, πολίτες μάλλον επιθυμούν. Άρα λοιπόν τι πρέπει να πούμε. Χρειάζεται περισσότερο συντονισμός. Αλλά περισσότερο συντονισμός σημαίνει επίσης νομιμότητα σε όλα αυτά. Και ο μόνος χώρος ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα όπου η νομιμότητα προέρχεται από τους ίδιους τους πολίτες ε, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά την άποψή μου δεν είναι θεμητό να σκεφτούμε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς τους μηχανισμούς χωρίς να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχοντας τις πολιτικές που θα αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι δικό σας καθήκον και έργο. Για να γίνει τώρα κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται να αλλάξει η συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχει ένα καλό μέσο, ένα εργαλείο στη συνθήκη, το 294, η φυσιολογική νομοθετική διαδικασία η, επιτρέπει τη συναπόφαση προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν και έγκριση αυτών από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι, αυτός είναι αυτοκινητόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε για περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο στην Ευρώπη και για να δοθεί δημοκρατική νομιμότητα, νομιμοποίηση σε δεσμευτικές νομοθεσίες. Εγώ στο έγγραφο προς την Επιτροπή σας έχω, γράψει στο δεύτερο τμήμα του πώς αυτές οι γενικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν μέσω πολύ συγκεκριμένων πολιτικών για τα θέματα που είναι επιτάπητος. Δηλαδή, ανταγωνιστικότητα, ανισορροπίες, ε, συντονισμός δημοσιονομικών πολιτικών και διαχείριση κρίσεων. Εγώ θα είμαι σύντομος. Για το πρώτο σημείο, την ανταγωνιστικότητα, είναι μια πολύ συγκεχημένη ιδέα. Ο Πολ μια φορά έγραψε ένα περίφημο άρθρο γι' αυτό. Και δυστυχώς η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, όλο ένα και περισσότερο εστιάζει τι ανισορροπίε των τρεχών του λογαριασμών, λε και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Αυτό είναι όμω λάθο. Μπορεί να υπάρχουν ε, καλές ανισορροπίες στους τρέχοντες λογαριασμούς και κακές. Οι καλές είναι η συνέπεια της ανάπτυξης, ε, της, ε, των, της οικονομικής δυναμικής και οι άσχημες είναι αυτές που σχετίζονται με την απώλεια ανταγωνιστικότητα τιμών και, και άλλων επίσης πραγμάτων. Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται με το κόστος της μοναδιαίο κόστος του εργατικού δυναμικού και αυτό σχετίζεται με την παραγωγικότητα. Και πάλι, Και αυτό ήταν πάντα ταμπού ανάμεσα στους υπευθύνοντες για τις πολιτικές αποφάσεις στην Ευρώπη. Το 1999 ο διάλογο μακροοικονομικής πολιτική δημιουργήθηκε ώστε να συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι σε ένα διάλογο με τι δημοσιονομικέ αρχέ και την Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι ένα κρυφό εργαλείο συντονισμού το οποίο δεν ξέρει κανείς τι κάνει. Και οι αρχές που έχουν συζητηθεί εκεί ποτέ δεν έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένες ε, ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις περί μισθών. Περισσότερο εστιαζόμαστε σε μη εμπορικού τομεί και ιδιαίτερα βόρεια στη Γερμανία στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Αυτό που θα ήταν σημαντικό είναι να ανοίξει αυτή η συζήτηση και να δημιουργηθεί διαφάνεια στην Ευρώπη, έτσι ώστε ως οι διαπραγματευόμενοι περιμισθών και οι σχετικές συζητήσεις στα ΜΜΕ να εξετάσουν το θέμα των αμοιβών ως ε, μια γενική ε, ένα γενικό προβληματισμό. Δεν χρειάζεται για να γίνουν νόμοι, ίσως ε, μόνο σε κάποιες ε, ειδικέ περιπτώσεις, αλλά χρειάζεται διαφάνεια. Και γι' αυτό και προτείνω ο μακροοικονομικός διάλογος να πάει από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να σχετιστεί με τις συζητήσεις που έχετε εσείς εδώ σε αυτήν την Επιτροπή πριν να γίνουν οι ακροάσεις με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεύτερον, σε σχέση με την δημοσιονομική πολιτική, περισσότερος συντονισμός προφανώς χρειάζεται, όμως αυτός ο συντονισμός των πολιτικών θα πρέπει να συνδυάσει την λιτότητα, την αυστηρότητα και την ευελιξία. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Ο Βενισμάκη είπε πριν από λίγο ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο προπολογισμό ε, στην ε, Ευρώπη και φυσικά έχει δίκιο και κανείς δεν θέλει να υπάρξει κάτι τέτοιο. Όμως το 40-45% του ΑΕΠ στην Ευρώπη δαπανάται από τις ε, κυβερνήσεις των κρατών μελών και αυτό είναι σωστό γιατί έτσι είναι η κατανομή των δημοσίων αγαθών σε προτιμήσεις κυρίως ε, εθνικών ψηφοφόρων και πολιτών, στο εθνικό τους δηλαδή συμφέρον. Ε, ωστόσο υπάρχουν εξωτερικές σχέσεις όπως είδαμε που προκύπτουν από την κατανομή αυτή διότι ε, συγκεκριμένα κράτη-μέλη επιδιώκουν πολιτικές που μπορεί να έχουν ε, επιρροή σε άλλες χώρες όπως είδαμε την Ελλάδα και τη Γερμανία και άλλους και άρα λοιπόν είναι σημαντικό να εσωτερικευθούν αυτές οι εξωτερικές ε, σχέσεις καθορίζοντας μια ομαδοποιημένη ε, δημοσιονομική πολιτική στάση για την Ευρωζώνη. Για την Ευρωζώνη είναι το πιο σημαντικό, για τις υπόλοιπες χώρες είναι λιγότερο επίγον. Τώρα, ο καθορισμός μιας συγκεκριμένης ε, στάσης για τη δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να εφαρμοστεί και πώς το εγγυόμαστε αυτό. Εγώ έχω κάνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση στο έγγραφό μου προς την Επιτροπή σας. Η βασική ιδέα είναι να μετατραπεί ένα τμήμα των ισχυουσών διαδικασιών σε νομοθεσία μακροοικονομικού πλαισίου. Αυτή δεν είναι νέα ιδέα. Ο γαλλικός εθνικός περιπολογισμός βασίζεται σε μια τέτοια νομοθεσία για την μακροοικονομική πολιτική και τα υπάρχει διατησία ανάμεσα στα διάφορα υπουργεία και στην εφαρμογή των πολιτικών και στην Ιταλία υπάρχει το TPF που είναι ένα άλλο μέσο, εργαλείο μάλλον μακροοικονομικής πολιτικής. Πρότασή μου είναι ότι αυτός ο νόμος περί μακροοικονομικής πολιτικής θα αυξάνει, αυξάνει το ομαδοποιημένο έλλειμμα για την Ευρωζώνη Και αυτό, ανάλογα με το ΑΕΠ, μπορεί αυτό να το τροποποιήσουμε, ας πούμε, λιγότερο σε εκείνους που έχουν υψηλότερο επίπεδο χρέους από ότι σε εκείνους που έχουν χαμηλότερο χρέος, έτσι ώστε με μονομένες χώρες μέλη να μπορούν να δανείζονται σε αντιστοιχεία με αυτά τα ποσά. Αυτό, αυτές οι άδειε επίσης θα μπορούν να μεταφερθούν. Δηλαδή δίνουν δικαιώματα δεν είναι μια ένωση ε, μεταφορών ε, με την έννοια ότι η μία χώρα δίνει στην άλλη, αλλά τα δικαιώματα μπορούν να μεταφέρονται. Να είναι δηλαδή ε, άδειες που θα μπορούν να μεταφερθούν όπως οι άδειες για την ρήπανση για παράδειγμα. Αυτό θα μπορεί να γίνει δηλαδή αν κάποια χώρα δεν θέλει να δαπανίσει και να δανειστεί τόσο πολύ, να το δώσει το δικαίωμά τη σε μια άλλη. Αλλά το σύνολο να διατηρείται. Το σύνολο ελλείμματο να διατηρείται σύμφωνα με τον, οικονομικό, με τον επιχειρηματικό κύκλο ή το οικονομικό κλίμα. Και αυτό οδηγεί σε έναν πολύ απλό μηχανισμό για την εφαρμογή όλων αυτών. Γιατί αν υπάρχουν άδειε δανεισμού, μπορεί κανεί να περάσει νόμου που θα λέει, ναι, ότι οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να δίνουν χρήματα μόνο στις δημόσιες αρχές, μόνο αν μπορούν να παρουσιάσουν τα αντίστοιχα ποσά σε αδίες δανεισμού. Αν μια κυβέρνηση δηλαδή δεν έχει άλλη άδεια, δεν μπορεί να δανειστεί άλλο. Και αυτός είναι ένας απλός τρόπος για την αποκεντροποίηση της εφαρμογής των δημοσιονομικών περιορισμών που είναι απαραίτητο, απαραίτητη, ενώ ταυτόχρονα δίνεται επαρκής ευελιξία. Επίσης, προσθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση, διότι προέρχεται από ένα νόμο πλαίσιο που έχει την πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τρίτο στοιχείο, διαχείριση κρίσης. Να σύντομος. Ανέφερα προηγουμένως στο Κοινοβούλιο την ιδέα, παλιότερα μάλλον στο Κοινοβούλιο, την ιδέα της έκδοσης ε, ομολόγων της Ένωσης, πράγμα το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που συζητήθηκε πριν εδώ με τον Επίτροπο, αλλά έχει σχέση με το τη διαχείριση των κρίσεων και βέβαια όλοι οι θεσμοί αγγίζουν το θέμα και είναι το θέμα του ηθικού κινδύνου. Και με αυτό θα θέλω, θέλω να ολοκληρώσω ως ένα θέμα αρχής. Ο ηθικός κίνδυνος είναι μια λειτουργία κανόνων και ανεξάρτητων φορέων. Με άλλα λόγια, υπάρχει ο ηθικός κίνδυνος μόνο επειδή υπάρχει ένας κανόνας και μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα κάνουν οι άλλοι σύμφωνα ανάλογα με τον κανόνα και προσπαθεί να το παρακάψει στην συνέχεια. Αλλά το θέμα του να υπάρχει όμως οικονομική, ε, του να υπάρχουν κυβερνήσεις είναι ότι οι κυβερνήσεις λειτουργούν διακριτικά και όχι μόνο υποκανόνες. Θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε τον ηθικό κίνδυνο εάν έχουμε μια σωστά εγκαθιδρυμένη δημοκρατική κυβέρνηση για τα οικονομικά ζητήματα που θα έχει απόλυτη νομιμοποίηση μέσω της δημοκρατικής διαδικασίας και έγκριση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτό θα γινόταν ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Θα μπορούσε δηλαδή η Κομισιόν να λάβει μέτρα με την απαραίτητη διακριτική ευχαίρεια ανάλογα με την περίπτωση δεδομένη τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε δημοκρατική διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο νομίζω πω η Ευρώπη θα έχει βρει τον τρόπο να προχωρήσει και θα ήταν μια μικρή δημοκρατική επανάσταση μέσα στο πλαίσιο της ε, συνθήκης της Λισαβόνα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμεί. και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αντρέ Σαπίρ ο οποίος είναι καθηγητής ε, οικονομικών ε, στο Μπρούγκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, όπως θα έχετε ίσως δει από τις δημοσιεύσεις μου, πάρα πολλά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν, ε, με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τη δική μου τη χρειά σε αυτή τη συζήτηση που αφορά στην ε, νομιμοποίηση, που συμφωνώ μαζί σας, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τι μάθημα μπορούμε να εξάγουμε από την κρίση για θέματα διακυβέρνησης. Τα μαθήματα που μπορούμε να εξάγουμε αφορούν την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων. Και θα μιλήσω κυρίως για την πρόληψη των κρίσεων, αλλά αν μου το επιτρέπει ο χρόνος θα ήθελα στο τέλος να πω και μερικά πράγματα για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρόληψη των κρίσεων και με το σύστημα εποπτείας. Το βασικό μάθημα που εξάγω από την κρίση είναι ότι πράγματι υπήρξε ανεπάρκεια. Ανεπάρκεια σε επίπεδο πειθαρχία αλλά και σε επίπεδο εποπτείας. Ανεπάρκεια προφανώς δεν υπήρξε μόνο σε εθνικό επίπεδο υπήρξε ανεπάρκεια και σε επίπεδο ευρωζώνης. Το παράδοξο της όλης ιστορίας είναι ότι σε εθνικό επίπεδο πράγματι δεν υπήρχε απαραίτητη κυριαρχία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή βλέπουμε υπουργούς που συναντώνται στις Βρυξέλλες, ε, ε, συναντώνται σε επίπεδο Eurogroup ε, πριν κατόπιν συναντηθούν σε επίπεδο ECOFIN και αυτά που συζητώνται σε αυτά, σε αυτά όλα τα συμβούλια δεν διαχέονται στα κράτη-μέλη. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ε, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις από αυτού, το σύμφωνο αυτό έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Η βασικότερη έλλειψή του είναι ότι τα κράτη-μέλη καλούνται ως κυρίαρχα να αντιμετωπίσουν τα δημοσιονομικά τους. Για δέστε λιγάκι την κατάσταση των διαφόρων κρατών. Αυτό το οποίο δεν κατόρθωσαν να πράξουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι να έχουν μία προσέγγιση εποπτείας μεμονωμένων κρατών μέσα από την ανάλυση των επιπτώσεων που θα είχαν οι πολιτικές τους στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι χώρες οι οποίες ε, σε εισαγωγικά συμπεριφέρθηκαν λανθασμένα ε, πράγματι ε, οι συνέπειες των πράξεών τους έγιναν ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η συζήτηση ποτέ δεν έγινε σε επίπεδο εποπτείας. Ε, συζητιόταν μόνο και λεγόταν ότι οι χώρες πρέπει να τηρούν τους κανόνες απλά και μόνο εξετάζοντας τα δικά τους, ε, τα στενά οικονομικά, όχι το ενδεχόμενο των επιπτώσεων στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Άρα δηλαδή καταλήγω στο ότι αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι ότι χρειαζόμαστε λιγότερη, αλλά διαφορετική εποπτεία. Κατά την άποψή μου, αυτό που πρέπει να έχουμε είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας. Το θέμα, παρότι συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, που στήριξε και ο κύριος Κοταρέλη και άλλοι που λένε ότι ε, θα πρέπει να έχουμε εποπτεία σε εθνικό επίπεδο εθνικοί δημοσιονομικοί κανόνες και δημοσιονομικές αρχές. Αυτό είναι κάτι ε, που μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ είμαι σαφώς ε, περισσότερο υπέρ των δημοσιονομικών αρχών, αλλά και αρχές αυτές θα πρέπει να είναι αρχές εποπτείας ε, των κανόνων. Δεν υπάρχει αντίφαση και διάσταση μεταξύ των δύο. Προφανώς υπέρ των ανεξάρτητων δημοσιονομικών αρχών, αλλά εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και μία ανεξάρτητη αρχή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωζώνης. Οι εθνικές λοιπόν αρχές και οι κοινοτικές ή ε, οι αρχές της Ευρωζώνης αυτοί όλοι θα πρέπει να αποτελούν αυτό που αποκαλούμε Ευρωπαϊκό Σύστημα Εποπτείας. Κατά την άποψή μου λοιπόν Εάν θέλουμε να έχουμε αυτό το σύστημα εποπτείας, και θα σας πω ευθύ αμέσω ε, με περισσότερη λεπτομέρειε τι εννοώ, να έχουμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο αποδίδει μεγάλη σημασία στην διατήρηση του κοινού αγαθού που είναι η Ευρωζώνη. Η έμφαση να δίδεται στην εποπτεία και όχι στα μεμονωμένα κράτη-μέλη, αλλά στο τι ακριβώς συνεπάγεται η συμπεριφορά μεμονωμένων κρατών μαλλών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης κυρίως. Νομίζω ότι ε, από όλα αυτά εξάγουμε το συμπέρασμα ότι εδώ χρειαζόμαστε νομιμοποίηση και αυτή είναι η νομιμοποίηση που εγώ είναι διαφορετική. Είναι νομιμοποίηση που προέρχεται από την εποπτεία η οποία έχει ως στόχο τη διαφύλαξη του κοινού αγαθού. Ένα σύστημα εποπτείας που αποτελείται από εθνικές ανεξάρτητες αρχές όπως είπαμε και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής οι οποίες ε, πρικοδοτούνται με μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Θα πάω τώρα στο ρόλο των εθνικών αρχών που είναι κάτι πολύ πιο εύκολο. Ας δούμε λιγάκι ποιος είναι ο ρόλος της ε, Επιτροπής των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμών. Προφανώς πολύ σημαντικός ο ρόλος του, του Eurogroup ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά κατά την άποψή μου το κομβικό στοιχείο στη νομιμοποίηση απορρέει από την ποιότητα της εποπτείας. Αυτό πρέπει να γίνει πάνω απ' όλα. Όσο η εποπτεία δεν είναι καλής ποιότητας, δεν είναι τέτοια που να αναγνωρίζει ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη, αυτό εννοώ εποπτεία καλής ποιότητας, αν δεν υπάρχει αυτό δεν θα κάνουμε, σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα της νομιμοποίησης. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να αρχίσουμε αναγνωρίζοντας κάτι επώδυνο, κάτι που όλοι μας περισσότεροι γνωρίζουν. Ότι τα προβλήματα που βιώσαμε την Άνοιξη αυτά σε μεγάλο βαθμό δεν είναι προβλήματα που απορρέουν από κακή συμπεριφορά μεμονωμένων κρατών. Η Ελλάδα τώρα βέβαια είναι μια ειδική περίπτωση. Η Ελλάδα είναι ειδική περίπτωση, αλλά δεν νομίζω ότι η Ισπανία, η Πορτογαλία η Ιρλανδία που αυτές είναι τελικά οι χώρες που προκάλεσαν την κρίση στην Ευρωζώνη. Ε, να μην ε, κάνουμε λάθη τώρα, αν το μόνο πρόβλημα ήταν η Ελλάδα, δεν θα αντιμετωπίζαμε την κρίση που βιώσαμε. Ας είμαστε ειλικρινείς. Άρα δηλαδή, Σήμερα μιλάμε για κυρώσει. Και αν υπήρχαν κυρώσει, τα προβλήματα ε, θα είχαν εξαφανιστεί. Δεν θα υπήρχε καν πρόβλημα, λένε μερικοί. Αυτό είναι πολύ απλουστευμένο. Αυτό ε, αποδίδει ιδιαίτερε ευθύνε στη συμπεριφορά μεμονωμένων κρατών, αγνοώντας όμως ε, τι επιπτώσεις στην Ευρωζώνη. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίσουμε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα εποπτείας Τη Ευρωζώνης. Όχι στο σύστημα εποπτείας μεμονωμένων κρατών. Γενικότερα, στο σύνολο εποπτείας στην Ευρωζώνη. Και αν το δούμε έτσι το θέμα, όλα αυτά περιλαμβάνουν και τη Γερμανία. Και δεν μπορούμε να εξετάζουμε την Ισπανία αγνοώντας τη Γερμανία. Δεν αποφαίνομαι το ότι η Ισπανία φερει μόνη το βάρος την ευθύνη ούτε η Γερμανία. Εγώ λέω η Ευρωζώνη το φέρει. Φέρει την ευθύνη. Άρα δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα εποπτείας που να εντοπίζει τα προβλήματα που πλήττουν την Ευρωζώνη και βεβαίως τη διάστασή τους σε επίπεδο κράτους μέλους. Αλλά δεν μπορούμε την εποπτεία να τη σχετίζουμε με μεμονωμένα κράτη αγνοώντας ότι αυτά ανήκουν σε μία Ευρωζώνη. Αυτό ισχυρίζομαι. Δεν λέω ότι δεν πρέπει κανείς να εξετάζει την κατάσταση μεμονωμένων κρατών και προφανώς ε, σε τελική ανάλυση ε, οι μοχλοί που πρέπει να κινητοποιηθούν είναι σε εθνικό επίπεδο. Αλλά εκείνο που λέω είναι να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στην Ευρωζώνη. Και μόνο έτσι μπορεί κανείς να κάνει συστάσεις σε μεμονωμένα κρατημέλη, ξεκινώντας από αυτή την σφαιρική αποτίμηση. Ε, Κατά τη δική μου άποψη, αυτή η μορφή εποπτείας είναι νόμιμοποιημένη για το ε, κοινό καλό της Ευρωζώνης. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σε επίπεδο αρχή είμαι κατά των κυρώσεων. Ε, αυτό είναι πολύ απλουστευμένο. Είναι σαν να λέμε κάποια κράτη συμπεριφέρθηκαν λάθος αντί να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα όπου όλοι μας και εγώ προσωπικά ε, και εγώ φέρω ευθύνη και εγώ δεν ε, διέβλεψα σωστά ορισμένα πράγματα. Αλλά το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Όλο αυτό το θέμα με τις κυρώσεις προκαλεί την εντύπωση ότι αν είχαμε εφαρμόσει κυρώσεις, αν ήμασταν πιο σκληροί δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Την Ελλάδα την αφήνω κατά μέρα. γιατί ένα κομμάτι του ελληνικού προβλήματος ε, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Μπορούμε όμως να πούμε ότι η Ελλάδα, ε, συγγνώμη με συγχωρείτε, η Ισπανία, η Ιρλανδία ε, δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά με τους κανόνες. Ας μην κάνουμε λοιπόν λάθη. Αυτό είναι ο λόγος που εγώ είμαι κατά των κυρώσεων. Γιατί σας λέω, οι κυρώσεις είναι υπεραπλουστευμένη λύση. Και ένας άλλος λόγος γιατί με κατά των κυρώσεων που έχει σχέση με τον πρώτο. Νομίζω ότι όσον αφορά την ποιότητα της εποπτείας εκεί σημειώνουμε πρόοδο. Προχωράμε σε μια πιο ευφύ εποπτεία. Και τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Από πλευράς δημοσιονομικής αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στη βιωσιμότητα. Και επίση σημαίνει ότι πρέπει να διευρύνουμε την οικονομική βιωσιμότητα, να ξεφύγουμε από τον οικονομικό τομέα και να περάσουμε και σε άλλους τομείς. Μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα, πάρα πολύ ωραία. Όπως είπε μόλις τώρα ο Στέφαν, από στιγμή που αρχίζουμε να μιλάμε για αυτό που θα έπρεπε να μιλάμε, δηλαδή για αυτά τα οικονομικά θέματα μεγάλης κλίμακας, μιλάμε για δημοσιονομική βιωσιμότητα, μιλάμε για ανταγωνιστικότητα και εγώ ως οικονομολόγος πρέπει να σας ομολογήσω κάτι. Εγώ δεν έχω τα εργαλεία για να μπορώ να αποφασίσω με ακρίβεια τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν τα κράτη. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό αν, ας πούμε, αν με ρωτάγατε για το ε, έλλειμμα του συζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ή αν με ρωτάγατε για την ανταγωνιστικότητα, μα ποια ανταγωνιστικότητα, εγώ μπορώ να σας πω ότι ε, το τάδε ποσοστό είναι πολύ μεγάλη απόκληση ε, και μετά θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις. Πώς μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Δεν είμαι διαιτητής όπως αυτός μπορεί να το κάνει η Κομισιόν. Επίσης στο θέμα της μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις όταν δεν επικρατούν οι ίδιοι όροι για όλα τα κράτη. Αλλά στο θέμα ε, το δημοσιονομικό μπορούμε να μιλάμε για ε, επιβολή κυρώσεων γιατί βλέπουμε τι συνέβη με ορισμένες χώρες ε, που συμπεριφέρθηκαν λάθος. Και ποιο είναι το κρίσιμο σημείο, το 3, το 4% έλλειμμα, πλεόνασμα. Δεν ξέρω. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι μια ευφύ αξιολόγηση και να καταλήξουμε ότι πράγματι το σύστημα ενέχει προβλήματα και ε, θα πρέπει να επαγρυπνούμε ως προς αυτά τα προβλήματα. Επίσης, ε, η ηθική ηθικές, νομιμοποιημένες ηθικές αρχές ε, θα πρέπει να φέρουν ευθύνη. Εδώ μπαίνει λοιπόν η νομιμοποίηση. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει ε, προβλήματα. Όμως αυτά τα προβλήματα δεν θα αντιμετωπιστούν, αντιμετωπιστούν με κυρώσεις. Και υπάρχει κάτι το καθοριστικό. Είτε θα παραμείνουμε στους απλούς κανόνες, δηλαδή κριτήριο 3% έλλειμμα ή... Ε, 3% έλλειμμα του συζυγίου ε, τρεχουσών συναλλαγών. Ο κανόνας αυτός εμπαρθώσει του 3% και στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ευφυές σύστημα εποπτείας, μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις. Εγώ δεν το θέλω αυτό, αλλά στην περίπτωση αυτή βλέπω ότι οι κυρώσεις απορρέουν από πολύ απλούς κανόνες. Ε, και αυτό το λένε και πολλοί άλλοι, αυτό είναι και το ε, σύμφωνο σταθερότητα. Η ομορφιά όλου αυτού του συστήματος είναι ότι, ενέχει, ότι περιλαμβάνει έναν αριθμό. Ε, το σέβομαι αυτό. Εντάξει, τα σέβομαι όλα αυτά. Όχι ότι συμφωνώ. Σέβομαι αυτή την άποψη γιατί είναι συνεπής. Ε, που λέει, αν δεν σεβαστεί το 3% θα υποστείς κυρώσει. Τώρα, αν ξεφύγουμε και πάμε στην αξιολόγηση μια κατάσταση κάτι που είναι πολύ ευρύτερο, δεν λέμε κριτήριο 3% έλλειμμα, αλλά μιλάμε για δημοσιονομική βιωσιμότητα. Και αν μιλάμε για βιωσιμότητα μιας ζώνης από το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας, ούτε εγώ, αλλά ούτε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο νομίζω ότι έχουν αριθμούς που να λένε ότι στην ανταγωνιστικότητα, άμα δεν σεβαστείς αυτόν τον αριθμό, ε, θα υποστήσει το ποσοστό, θα υποστήσει κυρώσεις. Άρα δηλαδή ή θα έχουμε απλό σύστημα των κυρώσεων ή ένα πιο ευφυές σύστημα εποπτείας που είναι ευρύτερο που όμως τότε θα πρέπει ε, να έχουμε άλλο διαιτητή, όχι αυτόν ε, που βγάζει την κόκκινη την κίτρινη κάρτα. Ε, θα έχουμε την ηθική εκείνη αρχή που θα κάνει την αποτίμηση και θα λέει εδώ η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει πρόβλημα και πρέπει να αναζητηθεί η λύση. Και η λύση δεν αναζητείται σε επίπεδο μονομένων κρατών, πρώτα να γίνεται αποτίμηση του συνόλου της Ευρωζώνης. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε ακριβώς τα ίδια όπως και κατά παρελθόν. Απλά θα προσθέτουμε νέα κριτήρια. Μου είπαν ότι τελειώνει ο χρόνος μου. Τέλειωσε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Προεδρεύων. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Σαπίρ και τώρα Έχετε τη δυνατότητα να θέσετε ερωτήματα, να κάνετε σχόλια. Ο κύριος Λάμπερτ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Τα σχόλια μου απευθύνονται στον Αντρέ Σαπίρ. Νομίζω ότι είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα όταν λέει ότι δεν μπορεί κανείς να κοιτάζει μόναχα μια χώρα μεμονωμένα. Πρέπει <clears throat> να δει κανείς τη χώρα σε σχέση με την σύνολη περιοχή του ευρώ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο στην περίπτωση αυτή. Αλλά εγώ θα έπαιρνα ένα διαφορετικό παράδειγμα από αυτό που διαλέξατε εσείς. Όταν μια χώρα όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία έχουν δημοσιονομικές πολιτικές, πολιτικές φορολογίες που βλάπτουν τις ίδιες τις χώρες αυτές γιατί δημιουργούν φυσαλίδες και άλλες χώρες επίσης βλάπτουν γιατί δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό και απορροφούν χρήσιμο κεφάλαιο για στόχους οι οποίοι δεν είναι παραγωγικοί, τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχετε δίκιο στο σημείο αυτό. Αλλά <clears throat> αλλά τελικά όλα αυτά είναι ουσιαστικά μία μεμονωμένη δράση καταχρηστική των χωρών αυτών. Όταν βλέπω την Ελλάδα να δαπανά 3 ή 4% του ΑΕΠ της σε άμυνα, σε αμυντικούς εξοπλισμούς, αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν είναι υγιές. Αν δείτε λοιπόν τι κάνουν χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, οι χώρες σαν τη δική μου, που κατά κάποιο τρόπο δημιουργούν μικρούς φορολογικούς παραδείσους, όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> και πρέπει να υπάρχει μια κύρωση, θα πρέπει να υπάρχει απειλή συνεπειών. Αυτή τη στιγμή ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Θέλει να κάνει κάτι το βέλιο με το φορολογικό του σύστημα, το οποίο ουσιαστικά θα αφαιρέσει φορολογικά έσοδα τη Σουηδία. Μπορεί να το κάνει. Αυτό δεν πρόκειται να το τιμωρήσει κανένα. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πιο ευφύς για τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε αυτά τα συστήματα να λειτουργήσουν. Αλλά μέχρι να έχουμε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση, η οποία είναι υπόλογη προς τους Ευρωπαίους πολίτες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά έχουμε απλώ εθνικές κυβερνήσεις και οι εθνικές κυβερνήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκλογέων τους και προσπαθούν να ικανοποιήσουν αυτούς. <clears throat> και μετά χρησιμοποιούν τις Βρυξέλλες σαν τον κακό μπάτσο. Λένε, κοιτάξτε θέλω να σα ε, ικανοποιήσω αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί δεν με αφήνουν οι Βρυξέλλε. Αυτό δεν δημιουργεί ένα θετικό συνέστημα εναντί τη Ευρώπη. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων. Για το θέμα τώρα τη νομιμοποίηση, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο διαφωνώ μαζί σα. Έτσι που παρουσιάσατε την νομιμοποίηση είναι νομιμοποίηση σημαίνει καλή εποπτεία. Αυτή είναι για μένα μια τεχνοκρατική προσέγγιση, ένα τεχνοκρατικό ορισμό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η νομοποίηση προέρχεται μονάχα από του πολίτε, από το λαό. Μπορεί να είμαι παλαιομοδίτικο, αλλά σε κάποιο σημείο η νομοποίηση πρέπει να έχει δημοκρατικό χαρακτήρα. Πρέπει εμεί, οι εθνικέ κυβερνήσει η Κομισιόν να είναι υπόλογοι προ του εκλογείς και πολίτε. Είναι ο μόνο βιώσιμο τρόπο να εξασφαλίσουμε νομοποίηση είτε έχουμε καλού κανόνε ή κακού κανόνε. Όλα τα άλλα είναι ένα τεχνικό θέμα, δεν είναι ένα πολιτικό θέμα. Ευχαριστώ. Ο κ. Δομενίτη τώρα έχει το λόγο. Και μετά οι καθηγητές θα απαντήσουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πολλές ε, λαβές, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Εγώ προσωπικά, δεδομένου ότι έγιναν πολλές ε, παρομοιώσεις με το ποδόσφαιρο, αμφιβάλλω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συγκριθεί με έναν διαιτητή, όπως είπε πριν ο Επίτροπος Ρένα, αλλά, εν αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Η ερώτησή μου είναι πολύ απλή και αφορά τη χώρα μου. Ποια είναι η δική σας άποψη σε σχέση με την πρόταση που έκανε η Ιταλική κυβέρνηση ώστε να ξαναμπεί στα κριτήρια αξιολόγησης του χρέους της χώρας η ποσοτική και ποιοτική σύσταση του ίδιου του χρέους και η σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό χρέος των Ιταλικών οικογενειών. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο να απαντήσετε τα ερωτήματα αυτά τα οποία τέθησαν. Okay, I will, uh, will start briefly with this uh, question. Θα αντιμετωπίσω εν συντομία το ερώτημα αυτό και ίσως μπορώ να κάνω κάποια σχόλια για αυτά που είπαν οι άλλοι αξιότιμοι κύριοι για το θέμα αυτό. Για το θέμα του δημοσίου εναντί του ιδιωτικού χρέους αυτό είναι σημαντικό θέμα. Πρέπει να δούμε και το χρέος των οικοκυριών. Παράδειγμα τώρα, αν, το, αν σκάσει το λάστιχο στο αυτοκίνητό μου, το λάστιχο του δημοσίου τομέα, φυσικά είναι πιο δύσκολο με δύο σκασμένα λάστιχα παρά μόνο με ένα σκασμένο λάστιχο. Αλλά πρέπει να δω, το γεγονός ότι πρέπει να δω και το άλλο λάστιχο το ιδιωτικό λάστιχο δεν σημαίνει ότι δεν είναι πρόβλημα να έχει κανείς ε, ένα λάστιχο το οποίο είναι σκασμένο και αυτό εμποδίζει το αυτοκίνητο να κινηθεί. Λοιπόν, για τα ζητήματα των χειρώσεων, αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι όχι τόσο το ενδιαφέρον των οικονομικών χειρώσεων, αλλά το θέμα των συνεπειών και του επιμερισμού των ευθυνών στις διάφορες χώρες. Κάτι το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα στην ζώνη του ευρώ σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Περίπου 2,6% του ΑΕΠ είναι το έλλειμμα στην περιοχή του ευρώ. Το μισό από ό,τι στις ΗΠΑ. Το πρωτογενές λοιπόν έλλειμμα, το συνολικό κρέος και η αύξηση του χρέους, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι δείκτες στην περιοχή του ευρώ είναι πολύ καλύτερα από τις Πολιτείες και την Ιαπωνία. Αλλά ανησυχούν οι χρηματαγορές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι οι άλλες περιοχές. Και παρόλα αυτά τα, ε, τα επιτόκια στην περιοχή του ευρώ και τα σπρέτς είναι πιο μεγάλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως έχει κάποια σημασία η σύνθεση του χρέους και ο ρόλος των μεμονωμένων κρατών μελών επίσης παίζει κάποιο ρόλο. Υπάρχει ίσως μια απλή, ίσως απλοϊκή αντιμετώπιση, αλλά υπάρχει το θέμα αυτό της ευθύνης, το οποίο είναι σημαντικό για όλους ε, στην καθημερινή ζωή. Αν οδηγώ ένα αυτοκίνητο και ξεπερνάω το όριο ταχύτητος, μπορεί να έχω το καλύτερο σύστημα παρακολούθησης, μπορεί να έχω ραντάρ, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αλλά δεν μου δώσει κανένα πρόστιμο όταν ξεπερνάω το όριο ταχύτητος, κανείς δεν πρόκειται να σέβεται τα όρια ταχύτητος. <clears throat> Νομίζω ότι η λογική του 3% είναι χρήσιμη αφέ αυτής, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την διχοτομική αντιμετώπιση ή έχετε ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ απλό ή κάτι το οποίο έχει διακριτικό χαρακτήρα και δεν έχει συνέπειες όταν κανείς κάνει παραβίαση των κανόνων. Να ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε το 2003, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Κολινιό. Ίσως να πρέπει να ξεκινήσουμε στο θέμα της σύνθεσης των δημοσίων δαπανών και τον ορισμό του τι ακριβώς είναι το, το έλλειμμα. Καταλαβαίνω γιατί η Ιταλική κυβέρνηση έχει κάνει μια τέτοια πρόταση θέλουν φυσικά να μειώσουν τους πιέσεις και τους περιορισμούς τους οποίους υφίστανται. Τώρα το θέμα είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε πώς η σύνθεση των δημοσίων δαπανών επηρεάζει την οικονομική απόδοση ή την οικονομική μεγέθυνση. Παρά το γεγονός ότι διαστητικά αυτό που λέτε είναι θετικό και χρήσιμο, από πρακτική έποψη δεν είναι χρήσιμο, δεν μπορεί να είναι εργαλείο δεν είναι εργαλείο να πετύχουμε τους πολιτικούς στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Για το θέμα του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, <clears throat> επίσης, πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορούν να υπάρχουν, όχι κατά ανάγκη, συμπληρωματικότητες μεταξύ των δύο. Αν δείτε την Ιαπωνία, έχουν γίνει μελέτες σε σχέση με την μακρά κρίση που μαστίζει την Ιαπωνία, η οποία φυσικά οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα χρέους έναντι ΑΕΠ στην Ιαπωνία. Επιχειρηματολόγησαν ορισμένοι επίσης ότι το γεγονό ότι η Ιαπωνική κυβέρνηση δανείζεται ενώ ο ιδιωτικό τομέα τα νοικοκυριά αποπληρώναν το χρέο του ότι μόνο αυτό έχει επιτρέψει στην Ιαπωνία να μην χρεοκοπήσει. Και ίσως αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο διαφορετική ίσως είναι διαφορετικές διαστάσεις σε σχέση με αυτό το οποίο βλέπουμε στην Ευρώπη. Αυτά μας οδηγούν σε ένα πιο σημαντικό ακόμα ερώτημα. Το ερώτημα αυτό είναι το εξή. Θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει μια σωστή πολιτική. Αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η σωστή πολιτική. Υπάρχει μια εσωτερική αντίφαση σε αυτά που λέει ο Αντρέα Σαπίρ. Λέει από τη μία πλευρά χρειαζόσαστε μια ανεξάρτητη δημοσιονομική αρχή. Πρέπει να είναι ένα σύστημα ανεξάρτητο, αλλά ανεξάρτητο από τι. Αυτό που είδαμε, αυτό το οποίο έχουμε δει να γίνεται κάθε μέρα στην Ευρώπη, είναι ότι οι ανεξάρτητες αρχές είναι απόμακρες, είναι απόμακρες και μπορούν να καταληθούν από συμφέροντα οικονομικά και πολιτικά και θεσμικά δεν ξέρουμε και ποια είναι η σωστή απάντηση. Μπορεί να υπάρχει μια συνένεση στις Βρυξέλλες όπως υπήρχε στη Ουάσιγκτον. Όπως λέει ο κ. Κοταρέλη, ότι σε σωρευτικό επίπεδο η θέση οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλύτερη από την των ΗΠΑ. Αλλά είναι καλό αυτό ή κακό, το ξέρουμε. <clears throat> Μήπως οι πολιτικές του Ομπάμα υποστηρίζουν περισσότερο την οικονομική ανάκαμψη και την επαναφορά της απασχόλησης στην παγκόσμια οικονομία από ό,τι κάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Τι ξέρουμε λοιπόν για όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό το οποίο θα να τονίσω είναι ότι αν νομίζουμε ότι έχουμε τις απαντήσεις επειδή είμαστε ανεξάρτητοι αρχή, τότε ουσιαστικά επικρατεί μία μονοκόμματη και μονολυθική σκέψη και η μονολυθική σκέψη οδηγεί σε αποτελέσματα που οι πολίτες μπορεί να μην τα ενσωματώνουν και να τα ενστερνίζονται όπως τους λένε οι τεχνοκρατικές αρχές. Επομένως, η νομοποίηση δεν προέρχεται από το να κάνουμε το σωστό από την ποιότητα. Η νομοποίηση συμ, συμ, προκύπτει και από την δημοκρατική συμμετοχή του, των πολιτών. Όχι μόνο αυτών που συμφωνούν, αλλά και αυτών οι οποίοι είναι αντιφρονούντες, που διαφωνούν. Αυτοί που μπορεί να έχουν τρελές ιδέες και διαμφισβητούν όλο αυτό το σύστημα. Και μετά πρέπει οι διαδικασίες αυτές, οι δημοκρατικές, να εξασφαλίσουν το ότι υπάρχει δημοποίηση, δηλαδή να υπάρχει αποδοχή από το λαό των πολιτικών οι οποίες αποφασίζονται. Δεν θα ήθελα να εμπλακούμε σε συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά δεν μπορώ και να αποφύγω τελείω τον πειρασμό. Δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να τοποθετηθώ σε αυτά που είπε ο κυρίος ε, Λαμπέρ. Ε, να πω κάτι σχετικά με αυτά που ελέγχθησαν. Που τα κατανοώ και που σε κάποιο βαθμό τα συμμερίζομαι Συμφωνώ ότι το θέμα της ε, νομιμοποίησης είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά και δύσκολο στην Ευρώπη. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Όμως, υπάρχει και ένα όμως. Προηγουμένως είπε ο Στέφαν ότι θα ήθελε να έχει ένα σύστημα όπου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωζώνης να είχαμε ένα συγκερασμό πολιτικών και να καταλήγαμε σε μία άποψη που κατόπιν θα διαχέεται στα κράτη-μέλη. Αλλά εγώ κάνω μια ερώτηση τους αριθμούς. Πού θα τους βρεις τους αριθμούς, τα στοιχεία για το ποιο είναι το επίπεδο ελλείμματος ή πλεονάσματος που χρειαζόμαστε για το σύνολο της Ευρωζώνης. Πώς θα το κάνουμε, θα το κάνουμε όπως ψηφίζουν στο Κοινοβούλιο, πώς θα καταλήξουμε στα απαραίτητα στοιχεία. Αυτά είναι δύσκολα θέματα. Ας πούμε, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συμφωνήσαμε να έχουμε μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εσείς αυτό το βρίσκετε λάθος. Εγώ δεν επιχειρηματολογώ υπέρ του να εκχωρήσουμε εξουσία σε ένα φορέα έτσι ώστε αυτός να μπορεί να καθορίσει το επίπεδο δαπανών, δημόσιων δαπανών ή εσόδων στην Ευρωζώνη. Εγώ λέω μόνο να υπάρχει μια ε, αρχή, ένας φορέας που θα αποφαίνεται, θα έχει άποψη και μετά θα ανοίγει η δημόσια συζήτηση. Δεν θέλω δηλαδή αυτός ο φορέας να σφετεριστεί την ε, εξουσία λήψη αποφάσεων. Το IMF να λέει την αδυσόπιτη αλήθεια. Όπως είπε και ο Κέινς. Θέλω λοιπόν να υπάρχει ένα σύστημα εποπτείας που θα περιλαμβάνει τόσο εθνικές αρχές όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρικοδοτημένα με μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Μεγαλύτερη ανεξαρτησία είναι μια προϋπόθεση που δεν αρκεί όμως. Μια άλλη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εποπτεία να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της ευρύτερης εποπτείας του συνόλου της Ευρωζώνης, όχι μεμονωμένων κρατών. Δεν πρέπει και να κοιτάει το κομμάτι, το κομματάκι της ντομάτας, το σύνολο, την ντομάτα της στρογγυλής, το σύνολό της. Κατ' ουσίαν λοιπόν μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν μιλάμε για κάποια θέματα φορολογίας, ε, τα οποία έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε άλλες χώρες φορολογικός ανταγωνισμός. Έχει αρνητικές επιπτώσεις. Ε, στην περίπτωση αυτή μιλάμε για τα ίδια θέματα όταν μιλάμε και για τις κρατικές ενισχύσεις. Δηλαδή μιλάμε για μέτρα που λαμβάνει μια χώρα εις βάρος της άλλης. Και αυτό είναι εύκολο να το κρίνει κανείς. Αλλά ε, δεν ήταν αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε την Άνοιξη. Το πρόβλημα ήταν ότι είχαμε πολιτικές οι οποίες κάποια στιγμή είχαν επιπτώσει σε όλους, όπως είπε και ο Λερέντσο και η Μάγκη. Και αυτό φοβόμαστε στην Ευρωζώνη. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν ήταν ελληνικό πρόβλημα, δεν ήταν ισπανικό. Φτάσαμε σε μια φάση όπου η βιωσιμότητα της ε, Ευρωζώνης ε, τίθετο σε κίνδυνο, ε, ε, διακυβεύεται. Αυτό έχει σημασία και αυτό εις βάρος του συνόλου της Ευρωζώνης. Άρα δηλαδή αν θέλετε εγώ κάνω αυτή τη διαφοροποίηση. Αυτά που είπατε εσείς για τον φορολογικό ανταγωνισμό, σε κάποια προϊόντα να έχουμε χαμηλή φορολογία, λυπάμαι καν... Εκείνο που συμβαίνει και συνέβη την άνοιξη στην Ευρωζώνη δεν ήταν ε, αυτό. Εκείνο που συνέβη ήταν ότι αμφισβητήθηκε η βιωσιμότητα του συνόλου της Ευρωζώνης. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει εποπτεία, διαφορετική εποπτεία στη ζώνη, κρίνοντας βέβαια και την πολιτική μεμονωμένων κρατών. Όμως ε, όπως σας είπα, έχοντας κατά νου το όραμα είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ο κύριος Λάμπερτ για να κάνει μια συμπληρωματική ερώτηση. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι για τα κριτήρια, για την εποπτεία και θέτω το ίδιο ερώτημα σε όλους τους ομιλητές. Μήπως θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια σε σχέση με την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων γιατί άμα χρησιμοποιεί κανείς μη ανανεώσιμους πόρους, αυτό είναι αρνητικό σε μακροοικονομικό επίπεδο και επίσης σε σχέση με δείκτες ανισότητες. Μπορεί να δει κανείς τις ανισότητες ότι είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που δεν λειτουργεί καλά, αλλά επίσης και σαν ένα χάντη κάποια την οικονομία. Θα θεωρούσατε λοιπόν ότι η χρήση ανανεωσίμων πόρων και η, το επίπεδο των ανισοτήτων είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια μορφή οικονομικής διακυβέρνησης. Τρεις συνάδελφοι ακόμα έχουν το λόγο, κύριο Πρεσέδο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Η οικονομική διακυβέρνηση είναι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Μια ένωση η οποία δεν πρέπει να είναι μονάχα νομισματική, αλλά επίση και οικονομική πολιτική. Ένωση οικονομική πολιτική. Αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι χρειαζόμαστε μια ευρύτερη σύλληψη όχι μονάχα η οικονομική πολιτική που είναι το άθροισμα της δράσης των 27 χωρών. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να υπάρξει οικονομικό συντονισμό χωρίς ένα γενικό οικονομικό πλαίσιο και χωρίς να σκεφτόμαστε το τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον Ευρωζώνης, ποιοι είναι οι στόχοι ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος είναι ο ρόλος της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να θεωρήσουμε ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες είναι να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν <clears throat> μπορεί πολλέ φορέ να μην ενισχύουμε τη θέση τη Ευρώπη στο διεθνές προσκήνιο. Επομένως και η εξωτερική διάσταση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι πολύ σημαντική. Πιστεύω επίσης ότι θα ήταν απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για την πολιτική μας, ενισχύοντας και τη θεσμική πτυχή, <clears throat> όχι μονάχα με την κοινοβουλευτική διάσταση, αλλά και κάποιες αρχές οι οποίες θα ενισχύσουν τον οικονομικό και νομισματικό πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις κυρώσεις. Εγώ έχω πολλές, ε, πολλούς δισταγμούς σε σχέση με τις κυρώσεις, ιδίως για τις αποδομητικού χαρακτήρα κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να καταστρέψουν κάτι το οποίο υπάρχει. αυτό το να κάνουμε κυρώσει μέσα σε μια εσωτερική αγορά που υποτίθεται δεν έχει κερδισμένου και χαμένου, αυτό δεν μπορεί να είναι υποφελέ. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε να έχουμε νέα εργαλεία και νέε ικανότητε μέσα στην οικονομική πολιτική και αυτό αφορά και το θέμα των ιδιών πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για να αντιμετωπίσουμε εξάλλου την κρίση, αυτό το οποίο πιστεύω ότι χρειάζεται είναι ένα ταμείο σταθερότητα, μονίμου χαρακτήρα, συζητήσαμε τη βοήθεια για ορισμένε χώρε υπό τον όρο οι χώρε αυτέ να έχουν να κάνουν επαρκή μέτρα, να πάρουν επαρκή μέτρα δημοσιονομικά. Αλλά κάποιε χώρε έχουν πιο γενναιόδωρα συστήματα κοινωνικά από ό,τι άλλε. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν μιλάμε για τον κοινωνικό χαρακτήρα τη οικονομία και για τον συντονισμό των οικονομιών. Κύριε Φιρέιρα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις. Οι ερωτήσει μου απευθύνονται κυρίω στον πρώτο μιλητή, γιατί κάπως με εξέπληξε το γεγονός ότι αναγνωρίσατε πως η Ευρωζώνη δεν έχει πρόβλημα ελλείμματο, δεν έχει πρόβλημα χρέους. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα της Ευρωζώνης? Γιατί ανησυχούμε, μα ανησυχεί τόσο πολύ αυτή η κατάσταση. Το πρόβλημα του Ευρωζώνη νομίζω ότι, από όσα είπατε, είναι το πρόβλημα των εσωτερικών διαφορών και ανισορροπιών. Και επειδή έχουμε το κοινωνόμισμα, αν ένα από τα κράτη-μέλη βγει εκτός προγράμματος, δημιουργείται ε, ε, πρόβλημα και στο υπόλοιπο σύστημα. Νομίζετε ότι η λύση γι' αυτό είναι κυρώσει. Εγώ ειλικρινά νομίζω πω δεν μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, αν η Ιρλανδία ή αν ε, η Ελλάδα ή οποιοδήποτε αντί να φτάνανε στο χρέο 80% ή 100% έπρεπε να δανειστεί λίγο περισσότερο για να πληρώσει την κύρωση θα βοηθούσε σε τίποτα, θα αποτελούσε αυτό κίνητρο για να συμμορφωθεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ παράξενο αυτό. Και αυτός ο μηχανισμός ήδη υπήρχε και δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Γιατί η Γαλλία ήταν μετά και η Γερμανία. Δεν θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει μέσα στην Ευρωζώνη. Γιατί το πρόβλημά μου όταν βλέπω την Ευρωζώνη είναι ότι ξεχνάμε το 3% και τα 60% ήταν μαζί σε συνδυασμό με μια πρόβλεψη ανάπτυξης για 3%. Σήμερα όμως αναπτυσσόμαστε, αρχίζουμε να αναπτυσσόμαστε για 1% και οι μακροπρόθεσμοι προοπτικές είναι 1%. Δεν είναι αυτό το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των αποκλήσεων στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη και επανέρχομαι στις παλιές ιδέες των ε, περιοχών συναγλωματικών ισοτιμιών. Δεν μπορείς να έχεις την ίδια εξωτερική πολιτική, το ίδιο νόμισμα, τα ίδια, την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία και τεράστιο ανταγωνισμό μέσα στην εσωτερική αγορά και μεγάλες αποκλήσει ε, στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα εντός ίδιου, του ίδιου χώρου χωρίς κανένα μηχανισμό για να το αντισταθμίζει αυτό. Γιατί η πολιτική συνοχής είναι κάτι το πολύ παλιωμοδίτικο με τον τρόπο που έχει φτιαχτεί είναι βασικά οι υποδομές. Και δεν το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Και ο προπολογισμό είναι πολύ μικρός. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα πιο σημαντικό από ότι οι κυρώσεις ή ένα κατάλογος, ένας κατάλογος κυρώσεων. Γιατί η απλότητα μπορεί να είναι όμορφη, αλλά υπάρχει ένα σωρό όμορφο κόσμο και ιδέε που δεν είναι μόνο ανόητε, αλλά και επικίνδυνε. Και εγώ βρίσκω ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ε, συμμετέχοντας είναι ο κύριος Κίγκολντ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι ανησυχώ λιγάκι για το πώς μπορεί να υπάρχει μια ευρεία συνένεση στο κοινοβούλιο μας τη στιγμή που ερχόμαστε από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και το είδα αυτό ήδη πριν που ήταν παρόντες οι δύο επίτροποι. Και επίση υπάρχουν διαφορές ύφους πολλές φορές μεταξύ μας που είναι αρκετά έντονες. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Για το κομβικό θέμα των κυρώσεων δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το κέριο θέμα ακόμα και οι εκλογείς που πιστεύουν στην αλληλεγγύη δεν δέχονται να δώσουν βοήθεια ή αντισταθμίσματα χωρίς την εγγύηση ότι κάποιες ενέργειες δεν θα επαναληφθούν. Θέλω όμως να προχωρήσω λίγο περισσότερο από αυτά που είπε ο κύριος Σαπίρ για το ερώτημα του πώς μπορούμε να διακριβώσουμε όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Στον τομέα του χρέους έχουμε κάποια συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, δεν υπάρχει παρά μόνο μια ασαφής οικονομική λογική πίσω από αυτά, δεν μπορεί κανείς να πει γιατί είναι 3 και όχι 4 ή 60 και όχι 80%. Τώρα το θέμα είναι γιατί βρεθήκαμε σε τέτοιες ε, δυσκολίες. Βρεθήκαμε σε δυσκολίες στις αγορές ε, αγαθών περιουσιακών, είχαμε εκρήξεις, φυσαλίδες ε, μεγέθησης στην αγορά ε, περιουσιακών στοιχείων, στα ακίνητα κυρίως και επίσης είχαμε και προβλήματα ανταγωνιστικότητας και εκεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μέτρο μέτρησης. Θα ήθελα να ξέρω αν οι άλλοι πανελιστές συμφωνούν με τον κύριο Σαπύρο ότι έχουμε πραγματικά προβλήματα καταμέτρησης, αν έχετε κάποιες ιδέες για το ποιοι είναι οι γνώμονες με τους οποίους μπορούμε να καθορίζουμε την ύπαρξη προβλημάτων ή όχι ουσιαστικά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί δεν έχουμε τελικά ένα σύνολο κανόνων το οποίο μπορεί να αποτρέψει ακόμα και τα είδη κρίσεων που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Αν λοιπόν είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, θα έχουμε τεράστια προβλήματα νομιμοποίησης, όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως. Θα ήθελα να αναφερθείτε λιγάκι περισσότερο στο θέμα του πώς μπορούμε <clears throat> να καταμετρήσουμε σωστά την έλλειψη ισορροπίας πέραν των καθαρών δημοσιονομικών δικτών. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω τώρα τους διακεκριμένους καθηγητές μας να απαντήσουν. Δεν χαίρομαι όμως πάρα πολύ. Γιατί συγχρόνως πρέπει να τους ζητήσω να παραμείνουν μέσα σε πέντε λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Κοταρέλη. Θα προσπαθήσω να μείνω στα πέντε λεπτά και θα ήθελα να Ξεκινήσω με αυτές τα μεγάλα ερωτήματα σε σχέση με τις δημοσιονομικές ανισορροπίες στο Ευρωζώνη. Ε, θα ήθελα να υποσαφηνήσω το εξής. Είναι σαφές ότι σε επίπεδο Ευρωζώνης το έλλειμμα είναι μεγάλο, είναι ψηλό. 6,5% είναι μεγάλο. Το, η αναλογία χρέους στην Ευρωζώνη ανάμεσα στο 2007 και 2015 θα αυξηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις μας κατά 25 ποσοστίες μονάδες. Δηλαδή δεν είναι μικρό το έλλειμμα λοιπόν και αυξάνεται και στην Ευρωζώνη, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο όσο στη ΣΥΠΑ. Αλλά τη δική μου θέση είναι ότι παρά το γεγονός, και εδώ έγκυται το πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι το έλλειμμα είναι μικρότερο, χαμηλότερο από ό,τι στη ΣΥΠΑ και στην Ιαπωνία, οι αγορές είναι πιο ανήσυχες για την Ευρώπη. Τα επιτόκια είναι ψηλότερα στην Ευρώπη από ό,τι στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Τα σπρέτζ είναι ψηλότερα κατά μέσο όρο από ό,τι στις είπα και στην Ιαπωνία. Υπάρχουν τώρα διάφοροι λόγοι στους οποίους οφείλονται όλα αυτά. Το ένα, ο σχετίζεται με την παρατήρησή σας, την ανάπτυξη. Δηλαδή, οι προοπτικές ανάπτυξη φαίνεται να είναι μεγαλύτερες για τη ΣΥΠΑ από ό,τι στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό, για παράδειγμα, εμείς είπα, εγώ έχω πει ότι το να σφίξει η δημοσιονομική πολιτική υπερβολικά πολλέ στην Ευρώπη θα είναι λάθος, γιατί αυτό μπορεί να σταματήσει την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν δημοσιονομικές προσαρμογές τουλάχιστον σίγουρα για τον επόμενο χρόνο, αλλά με προσοχή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προωθηθεί το δυναμικό ανάπτυξη στην Ευρώπη μέσω διευθυντικών αλλαγών. Αυτό είναι ένας λόγος. Ταυτόχρονα πιστεύω πως ε, υπάρχει η αντίληψη και είναι ε, βάσιμο αυτό ότι σε μια νομισματική ένωση οι πιο αδύναμοι κρίκοι είναι αυτοί που καθορίζουν την αδυναμία ολόκληρης αλυσίδας. Οπότε γι' αυτό η θέση των ε, πιο αδύναμων χωρών είναι πολύ σημαντική. Και όταν λέω για κυρώσεις, θέλω να αποσαφηνίσω και αν το ανέφερα αυτό και νωρίτερα, ότι μιλάμε για συνέπειες, για ε, επιπτώσεις της παράβασης κάποιων νόμων. Ε, Μπορεί να είναι και θετικέ επιπτώσει. Α πούμε, αν κάποιο συμπεριφερθεί σωστά, μπορεί να έχει πρόσβαση σε περαιτέρω πόρου από την κεντρική πηγή. Ε, ε, η βασική ιδέα ωστόσο ήταν ότι αυτό που πήγε στραβά, ξεκίνησε το 2000, από το 2003, ήταν ότι οι χώρες παραβίαζαν κάποιους κανόνες χωρίς να έχουν καμία επίπτωση. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Πρέπει να υπάρχουν κάποιε πτώσει για την ε, κακή συμπεριφορά και ανταμοιβέ για την καλή συμπεριφορά, αντίστοιχα. Για το θέμα το πώς ε, μετρώνται οι ανισορροπίες που δεν είναι δημοσιονομικές. Εγώ θα προχωρήσω ε, ο συνάδελφος εδώ που έλεγε ότι οι οικονομίες δεν έχουν κανένα εργαλείο κάτι το οποίο θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι η οικονομία δεν είναι η επιστήμη της τελειότητας, αλλά υπάρχουν πολλά μπορεί να πει κανείς για ορισμένες περιπτώσεις όπου το εξωτερικό χρέος είναι εξαιρετικά ψηλό ή όχι. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ίσως ε, θα ήταν άδικο να πούμε ότι υπάρχει ένας μόνο δείκτης που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει, αλλά δεν θα ε, πήγαινα τόσο μακριά ώστε να πω ότι δεν μπορεί να πει τίποτα για αυτά τα θέματα οικονομική επιστήμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Κολυνιό. Προηγουμένως σας είπα ότι ο ανταγωνισμός είναι μια συγκεχημένη έννοια και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποιοι πρέπει να είναι στόχοι μας για την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν δύο διαφορετικές έννοιες που έχουν σημασία στην συζήτηση στην Ευρώπη. Καταρχήν υπάρχει η γερμανική προσέγγιση στον ανταγωνισμό. Λέει να είμαστε αποδοτικοί, να είμαστε ε, σύγχρονοι, να έχουμε ένα προτέρημα εναντί των άλλων μέσω της τεχνικής και επομένως να καταλαμβάνουμε νέες αγορές. Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση στην ε, ε, ανταγωνιστικότητα που είναι να είναι κανείς φθηνός, να κερδίζει μερίδιο αγοράς, να μπορέσει να πλουτίζει σε βάρος των άλλων. Αυτό γίνεται και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ των δύο αυτό ενιών ή ιδεών δεν υπάρχει κοινό έδαφο. Δηλαδή, αν πάρει κανεί τη μία ή την άλλη άποψη, καταλήγει σε τελείω διαφορετικά συμπεράσματα σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα του Σφεν Χίγκολ για το πώ πρέπει να μετρήσουμε τι ανισότητε ή την ανταγωνιστικότητα. Εγώ δεν θέλω αυτό το, να συζητώ αυτό το επιχείρημα της ανισότητος σε ανταγωνιστικότητα γιατί προσπαθεί κάπως να συλλάβει την πραγματικότητα συλλήβδη. Υπάρχουν πολλά οικονομικά στοιχεία. Σε ορισμένε περιπτώσεις είναι καλό να υπάρχει έλλειψη ισορροπίας γιατί αυτό μπορεί να επιταχύνει την ανάκαμψη σε ορισμένε περιοχές. Μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις <clears throat> ισορροπιών σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές μεταφορές. Οι πλούσιοι πληρώνουν για τους φτωχούς. Αυτό είναι καλό. Αν επίσης μειώνται οι φόρες σε ορισμένε χώρες για να προσελκυστούν επενδύσεις, αυτό δεν είναι κακό κατά ανάγκη. Το θέμα είναι μέχρι που φτάνει κανείς. Βέβαια, οι, στοιχοί, οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων των ακινήτων παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τη Φλόριντα στην Νότια Ισπανία για να πηγαίνουν εκεί πέρα οι συνταξιούχοι Γερμανοί. Όλα αυτά είναι θέματα τιμών, κόστου στοιχείων που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο δεύτερο πυλώνα της πολιτικής παρακολούθησης της, εποπτείας, υπάρχει το θέμα του εμπορίου. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ εμπορίου μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξωτερικού εμπορίου. Βλέπετε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Η μόνη χώρα η οποία έχει αυξανόμενα πλεονάσματα και εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός είναι η Γερμανία. Όλες οι άλλες χώρες όμως που έχουν διαφορετικά ελλείμματα εδώ και δεκαετίες σε εσωτερικό και σε εξωτερικό εμπόριο δεν έχουν τόσο καλή θέση. Πρέπει να το δείτε λοιπόν αυτό συγκεκριμένα πώς γίνεται σε κάθε περίπτωση. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τελικά πρέπει να δούμε όλη την οικονομική πολιτική σαν ένα πακέτο. Πρέπει να το συζητήσουμε σαν σύνολο. Προφανώς έχεις δίκιο, υπάρχουν διάφορε απόψεων μέσα στην αίθουσα αυτή και μέσα στην Ευρώπη. Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. Αλλά η λογική τη δημοκρατία, όλα αυτά που έχουμε μάθει από την εποχή του Ancien Regime πριν από τη Γαλλική Επανάσταση όταν ήξερε μόνο ο βασιλιάς και ευγενιστή ήταν σωστό, είναι ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συνένωση με δοκιμέ και αποτυχίε, θα κάνουμε λάθη, θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα με την τωρινή θεσμική αρχιτεκτονική είναι ότι δεν έχουμε αρκετή ευκαμψία ότι οι συζητήσεις ουσιαστικά τις ε, απάγουν κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμένα συμφέροντα και ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταφέρνει να επιβάλλει τις προτιμήσεις τους σε όλους τους άλλους. Δεν έχουμε εργαλεία για να εξασφαλιστεί μια δημοκρατική απάντηση σε όλα αυτά τα θέματα και να μπορέσει κάποιο να πει ότι αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση ενδεχομένω. Μερικέ φορέ μπορεί να είναι και προ το συμφέρον τη Γερμανία να του πούν σκάστε και μην κάνετε αυτά που κάνετε. Και δεν ξέρετε εσεί όλη την αλήθεια. Και επομένω αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν οι δημοκρατικέ βάσει του πώ λειτουργεί η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τελευταίο για το ότι δεν πάει καλά με τις οικονομικές μα πολιτικέ. Δεν νομίζω ότι είναι μονάχα οι ανισορροπίες όπως είπα. Υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο ότι μέσα από μισό αιώνα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχουμε δημιουργήσει ορισμένα κοινά αγαθά τα οποία τα μοιράζονται όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες τα οποία είναι αλληλένθετα τα οποία επηρεάζουν και αφορούν όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα κοινά αγαθά χρειάζεται να τύχουν διαχείρισης και διακυβέρνηση με ένα συνεκτικό τρόπο. Αλλιώς δεν θα είμαστε στο βέλτιστο επίπεδο, αν θέλετε να το πω ακαδημαϊκά, θα είναι απλώς ολέθριο στην κανονική ανθρώπινη γλώσσα. Αν δεν έχουμε τη σωστή συνεκτικότητα, αν δεν εξασφαλίσουμε ότι όλες οι ενέργειες που κάνουμε προς μια κατεύθυνση ακολουθούνται από επαρκή συνεκτικότητα στο σύνολο, δεν θα έχουμε πετύχει. Κάναμε ένα βήμα τέτοιο με τη δημιουργία του ευρώ. Αλλά δεν έχουμε παρακολουθήσει με τις απαραίτητες διαδικασίες μακροοικονομικής διακυβέρνησης. Το πρόβλημα δεν είναι ότι κάποιες χώρες έχουν περισσότερο χρέος από άλλες. Κανείς μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι υπάρχει κάποιο κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο είναι αφαιρέγγιο, που δεν μπορεί να, ξέρει ξεπληρώσει το χρέο του, ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί πράγματι να πληρώσει στο μέλλον το χρέος του. Αυτό το οποίο έχουμε και το οποίο συνέβη φέτος ήταν μια κρίση ρευστότητα, όπου χώρε οι οποίες μακροχρόνια είναι βιώσιμε δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβαση στι αγορές γιατί οι αγορέ δεν του είχαν εμπιστοσύνη. Και όπω είπε ο Λορέντζο, οι αγορέ δεν έχουν πάντα δίκιο. Επομένως, χρειάζεστε ένα πλαίσιο για να παρέχεται ρευστότητα για τις κυβερνήσεις των κρατών μερών που έχουν προβλήματα πρόσβασης στις αγορές. Ήμουν τον Απρίλιο στο Πεκίνο στην αρχή της κρίσης και μίλησα με κάποιους εξέχοντες επενδυτικούς τραπεζίτες στην Κίνα που είπαν δεν θα αγοράσουμε τίποτα πια, κάνα περιουσιακό στοιχείο στην Ευρώπη γιατί δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κανένα δανειστή σε τελική, τελικής καταφύγης. Ξέρουμε πώς δουλεύει η, η Αμερικανική κυβέρνηση, ο Ομπάμα, η Αμερικανική Federal Reserve, θα αγοράσουμε δολάρια. Αλλά εάν εμεί δεν διορθώσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη, θα μας σβήσουν. Ο καθηγητή Σαπίρ. Σας ευχαριστώ. Για τον Κάρλο δεν ήθελα να πω ότι η οικονομική επιστήμη δεν μπορεί να πει τίποτα για τα θέματα αυτά. Τουλάχιστον δεν ήθελα αυτό να καταλάβετε. Αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορεί να πει ε, οτιδήποτε με αρκετή βεβαιότητα, ώστε να μπορέσουμε να το συνδέσουμε αυτό με αυτόματες κυρώσεις. Φυσικά και έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά ή θεωρώ ότι εγώ η κρίση μου είναι επαρκώς ασφαλής και βέβαιη ώστε να πω όχι, μέχρι εδώ και μη παρέκει και από εδώ και μπρος βάζω κυρώσεις. Όχι. Αυτό είναι που έλεγα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο που είπαμε ότι δεν συμφωνώ με τη γενική μας κρίση ή άποψη. Όχι, είπα ότι δεν είναι όλα αυτά απόλυτα βέβαια. Όποια είναι η αρχή που είναι υπεύθυνη εδώ, η δική μου ηθική αρχή, για μένα είναι η Κομισιόν εδώ, ας πάμε και ας πούμε υπάρχει πραγματικό πρόβλημα εδώ και ας ε, ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση. Τότε, αυτό είναι προτιμότερο από το να κρυφτούμε πίσω από αυτή την αυστηρή και απλουστευτική νομοστευτικό κανόνα που λέει ναι, έχει στάσει σε αυτό το σημείο και εδώ πρέπει να γίνει το εξή. Όχι, αυτό δεν λειτουργεί. σε κάποια φάση και θα είμαι σύντομος, δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί μιλάμε για νομιμοποίηση και είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Εγώ άλλαξα πολλές απόψεις για το τι συνέβη το 2003 με τη Γερμανία. Κατά κάποιο τρόπο η γερμανική κυβέρνηση υιοθέτησε την άποψη ότι Αυτά που θέλαν να, να κάνει η Κομισιόν δεν ήταν αποδεκτή. Δεν ήταν νομιμοποιημένο. Και υπονόμευσε ολόκληρο το σύστημα. Εγώ λοιπόν είχα δει πολλές και διάφορες απόψεις. Θα πρέπει να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να πούμε Αναρωτήθηκα λοιπόν, είναι, ήταν η Γερμανία τότε σε θέση δημοσιονομική που να θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη γερμανική βιωσιμότητα της δημόσιας οικονομίας της, αλλά τη βιωσιμότητα ολόκληρη της Ευρωζώνης. Ειλικρινά δεν μπορούσα να αποφασίσω. Άρα λοιπόν δεν, δεν ε, συμφωνούσα και τότε δούλευα στην Κομισιόν. Δεν συμφωνούσα με τη θέση της Κομισιόν που έλεγε ναι, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις στη Γερμανία. Γιατί ως οικονομολόγος εγώ δεν μπορούσα να καταλήξω σε αυτή την απόφαση. Να πω ναι, ότι η Γερμανία κάνει κάτι τρομερό και φοβερό τόσο για την ίδια όσο και για την Ευρωζώνη. Δεν μπορούσα να καταλήξω με βεβαιότητα σε αυτή την ε, κρίση. Από την άλλη πλευρά μπορούσα να δω ότι μέσω αυτής της συμπεριφοράς η Γερμανία που είχε ζητήσει το σύμφωνο σταθερότητας και που ήταν το ίδιο υπεύθυνο γιατί ήθελε να επιβάλλει δικαίως ή αδίκως ότι ήταν ε, η βάση της σταθερότητας ε, και ότι το ίδιο είχε αποδυναμωθεί και άρα επέφερε αστάθεια δεν, δεν έθετε σε κίνδυνο τα πάντα η Γερμανία μέσω τη οικονομική τη συμπεριφορά, αλλά λόγω τη πολιτική τη συμπεριφορά. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξει κανεί σε κάτι τέτοιο και κατά την άποψή μου δεν είναι πάρα πολύ θεμητό αυτό, δεν είναι πολύ νόμιμοποιημένο αν δεν μπορούμε δηλαδή να φτάσουμε στην καρδιά του ζήτηματο. Ποια ήταν η ουσία. Η ουσία δεν ήταν ότι η Γερμανία ε, ξεπερνούσε το 3%. Όχι, το, η ουσία ήταν ότι η Γερμανία ε, ε, ρισκάριζε να καταστρέψει ολόκληρο το σύστημα. Και γι' αυτό και η συζήτηση γινόταν σε ένα επίπεδο διαφορετικό από αυτό που έπρεπε. Γι' αυτό και αυτό, αυτό ζητώ, να μιλήσουμε για τα πραγματικά ζητήματα. Μην κρυφόμαστε πίσω από τους αριθμούς, γιατί αυτοί οι αριθμοί είναι δύσκολο να εξηγήσει στους πολίτες τι τους κάνεις. Αν υπήρχε πρόβλημα λοιπόν τότε έπρεπε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό απαιτεί η ηθική αρχή και ε, η ηγετική ικανότητα. Η ηθική αρχή είναι αυτή που έπρεπε να το σταματήσει. Ο κύριο Κοταρέλη θέλει να πει κάτι ακόμα. Ναι, θέλω να πω μόνο ότι σε αυτό συμφωνώ. Νομίζω ότι το θέμα των υπάρχει υπερβολικός αυτοματισμός με, βάση ένα συγκεκριμένο νούμερο ε, δεν είναι, είναι πολύ απλοποιημένη. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα συνδυασμός ε, νούμερων ε, ίσως το 2003 δεδομένων των συνθηκών η Γερμανία να μην δημιουργήσει πρόβλημα όσον αφορά τα νούμερα εκτός του ότι δεν θέτει σε κίνδυνο την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Γι' αυτό συμφωνούμε, από συμφωνούμε. Μάλιστα, πριν κλείσουμε αυτή τη δημόσια κρόαση θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους τρεις διακεκριμένους ομιλητές μας σήμερα και να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος Φανορομπόη έχει ένα μήνα μπροστά του για να παρουσιάσει την πρότασή του την πρόταση της Task Force για το πώς θα βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση και η σταθερότητα. Και θα έχουμε επιτάπητος πολύ ουσία για να κρίνουμε και να συζητήσουμε μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πολύ.